Αγαπητοί συνάδελφοι, καλησπέρα σας. Καθίστε παρακαλώ. I... I would like to... Θα ήθελα να σας καλωσορίσω όλους τους εκπροσώπους των Εθνικών Κοινοβουλίων, καθώς επίσης και τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην 29η έκδοση ε, της Ευρωπαϊκής Κοινοβουλευτικής Εβδομάδας. Θέλω να καλωσορίσω και την Κάρμεν Ελιάνα Μιχαλτσέσκου, αντιπρόεδρο ε, της Βουλής της Ρουμανίας, που θα συμπροεδρεύσει σε αυτό το πάνελ. Θέλω να ευχαριστήσω επ' ευκαιρία τη Ρουμανική Βουλή για τη στενή συνεργασία που έχουμε και είχαμε στη διοργάνωση αυτής της διάσκεψης. και χαίρομαι που σας βλέπω εδώ τόσο πολύ αριθμούς. Και σήμερα και αύριο θα έχουμε ένα διήμερο, πιστεύω, χρήσιμο και ενδιαφέρον ως ευκαιρία ανταλλαγής απόψεων ε, για την ευρωπαϊκή οικονομική διακυβέρνηση, την οικονομία γενικώ και τη βελτιωμένη συνεργασία μεταξύ των βουλευτών Εθνικών Κοινοβουλίων και Ευρωκοινοβουλίου. Σήμερα σε αυτή την αρχική σύνοδο θα ασχοληθούμε με το οικονομικό εξάμεινο και πώς έχει μέχρι σήμερα ε, λειτουργήσει στην πράξη. Ε, ερωτηματικό. Όπως γνωρίζετε το οικονομικό εξάμεινο είναι ένα πλαίσιο συντονισμού των εθνικών οικονομικών πολιτικών. Μια συνεχιζόμενη και διαρκής διακυβέρνηση και απάντηση, ε, όπως γνωρίζετε, ε, την ε, διαδικασία μακροοικονομικής σταθερότητας, ακολούθησε το σύμφωνο σταθερότητας και μετά ε, το ε, διπλό πακέτο, το TUPAC και στα τέλη του έτους, όπως γνωρίζετε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προτείνει μια, μια αναθεώρηση. Είναι μια καλή ευκαιρία λοιπόν να κάνουμε μια αποτύπωση της κατάστασης, μια αποτίμηση των εμπειριών είναι πολύ περίπλοκοι οι κανόνες όπως γνωρίζετε και όχι μόνο. Η αρμοδιότητα είναι αρμοδιότητα συντονισμού όπως ορίζεται από τη συνθήκη. Υπάρχει ένα νομικό πλαίσιο που είναι περισσότερο συγκεκριμένο σε κάποιους τομείς και λιγότερο συγκεκριμένο σε κάποιους άλλους. Πράγμα που έρχεται να ε, περιπλέξει έτσι περαιτέρω την κοινή μας διακυβέρνηση. Γι' αυτό λέμε ότι χρειάζεται βελτίωση. Ιδιαίτερα καθώς έχουμε και νομισματική ένωση και όχι μόνο ε, νέα αγορά. Όλα αυτά τα θέματα θα κυριαρχήσουν στη διάσκεψη. Ε, πριν αρχίσουμε όμως να σας πω κάποια οργανωτικά. Πώς θα ζητάτε το λόγο να τονίσω ότι κάνουμε ό,τι μπορούμε, όπως πάντα, έτσι ώστε να πάρουν το λόγο όσο γίνεται περισσότεροι συμμετέχοντες, ακόμα και σε περιορισμένο χρόνο, στον περιορισμένο χρόνο που έχουμε. Επειδή είναι πολλοί συμμετέχοντες, μετά από την εισαγωγή θα μιλήσετε, αλλά όχι σήμερα όλοι. Γι' αυτό σας παρακαλώ να περιορίζετε σε 2-3 λεπτά στην ε, παρέμβασή σας, θα βλέπετε και το χρονόμετρο και ανάλογα με τις συζητήσεις και την πορεία τους μπορεί να χρειαστεί και άλλη ένα προσαρμογή ο χρόνος. Θα βρείτε στα έδρανά σας κάποια δελτία που μπορείτε να συμπληρώσετε σε περίπτωση που θέλετε να πάρετε το λόγο και θα την παραδώσετε στους κλητήρες. Αυτό ισχύει και για τα μέλη των Εθνικών Κοινοβουλίων και για τους Ευρωβουλευτές. Γενικά θα προσπαθήσουμε να μοιράσουμε το χρόνο αγόρευσης έτσι με μια ισόρροπη φόρμουλα με ευελιξία. Και τώρα θα δώσω το λόγο και την Προεδρία στην κυρία Κάρμεν Λεάννα Μιχαλτσέσκου. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Γκουαλτιέρη. Είναι μεγάλη χαρά που συμπροεδρεύω μαζί σας ε, σε αυτήν την εκδήλωση. Από την άποψη της Ρουμανίας, αγαπητοί συνάδελφοι, η ενδυνάμωση ε, της συμμετοχής όλων σε αυτή τη διαδικασία είναι σημαντική έτσι ώστε να ενδυναμωθεί και ε, το ε, εξάμεινο και σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η Ρουμανία ε, που ασκεί την Προεδρία προσπαθεί να ε, ευθυγραμμίσει το εξάμεινο με τον οδικό χάρτη. Πιστεύουμε ότι το ευρωπαϊκό εξάμεινο παραμένει ένας πολύ καλός τρόπος συντονισμού των οικονομικών δραστηριοτήτων και στρατηγικών δεν έχουμε πολύ χρόνο, πρέπει να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας. Γι' αυτό λοιπόν ε, θα ήθελα να δώσω το λόγο στον πρώτο ομιλητή μας, μάλλον στην πρώτη ομιλήτρια. Στον πρώτο ομιλητή. Mr. Valdis. Στον πρώτο ομιλητή λοιπόν, τον κύριο Βάλτης Δομπρόφσκης, ε, χαίρομαι πολύ που είστε εδώ και που μπορώ να σας δώσω το λόγο. αξιότιμοι συμπρόεδροι, βουλευτές, κυρίες και κύριοι. Χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ σήμερα μαζί σας και που μπορούμε να συζητήσουμε για το Ευρωπαϊκό Εξάμενο. Το Ευρωπαϊκό Εξάμενο ε, είναι περίπου 10 ετών πλέον και έχει ε, δει και κάποιες ε, αλλαγές δίνοντας περισσότερο χώρο για τις εθνικές αρχές, τα εθνικά κοινοβούλια, εμπλεκόμενους, κοινωνικούς εταίρους κλπ. Ε, ήδη από πολύ νωρίς αναγνωρίστηκε το γεγονός ότι εξαρτάται η επιτυχία του εξαμήνου από κάποια στοιχεία. Πρώτον, η, η ποιοτική ανάλυση θα πρέπει να είναι το εξάμεινο αξιόπιστο και η αξιοπιστία ε, βασίζεται σε ε, σαφή ε, στοιχεία και αξιόπιστη ανάλυση επίσης ε, σημαίνει ότι θα πρέπει οπωσδήποτε η πραγματογνωμοσύνη να αντλείται από εσωτερικές και εξωτερικές πηγές. Το δεύτερο στοιχείο είναι η επικοινωνία. Ε, στις περισσότερες συστάσεις ε, δεν προβλέπονται ποινικέ κυρώσεις σε περίπτωση μη συμμόρφωσης. Άρα μιλάμε για ήπια εξουσία, soft power Πρέπει οπωσδήποτε, επομένως, να επικοινωνούμε τις αξιολογήσεις μας, οι οποίες θα πρέπει να γίνονται ορατές και γνωστές σε όλους τους εμπλεκομένους, κυρίως δε σε τους ε, βουλευτές, σε εθνικούς βουλευτές, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι και για την σχετική νομοθεσία. Ε, εμείς στην Κομισιόν συζητούμε συχνά ε, και τακτικά το εξάμεινο και με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και επιτόπου στις διάφορες χώρες χώρες, ε, ε, καθώς επίσης και με τους κοινωνικούς εταίρους. Ε, τέλος, τρίτο στοιχείο και πιο σημαντικό είναι η ιδιοκτησία, η οικειοποίηση. Αυτό συχνά σημαίνει ότι πρέπει κανείς να έρθει σε αντιπαράθεση με ισχυρά συμφέροντα, έτσι ώστε να υπερισχύσει εν τέλει το συμφέρον της χώρας. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να έχει υπάρξει ο μέγιστος βαθμός οικειοποίησης. Με τον τρόπο αυτό ε, και οι συστάσεις προχωρούν σωστά και τα κράτη ε, κάνουν τις, ε, τους απαραίτητους ελέγχους μέσω διαδικασίας ελέγχου από ομοτήμους και επισκοπήσεις. Βεβαίως μπορεί κανείς να αναρωτηθεί εάν όλα αυτά τα στοιχεία, τα τρία που ανέφερα προηγουμένως, εάν υπάρχουν, γιατί γιατί δεν υλοποιούνται όλες ε, οι συστάσεις. Αλλά αυτό ε, το ερώτημα θα ήταν υπερβολικά απλοϊκό, διότι εξορισμού ε, οι μεταρρυθμίσεις παίρνουν χρόνο. Γι' αυτό ε, λοιπόν είναι πιο λογικό να δούμε τα πράγματα σε πολυετή βάση έτσι ώστε ε, ο βαθμός υλοποίησης να είναι υψηλότερος. Όταν το 2014 ανέλαβε αυτή η Επιτροπή, 17 χώρες ε, βρίσκονται σε διαδικασίες υπερβολικού χρέους καθώς επίσης και υπερβολικής no Euro και υπερβολικού ελλείμματος. Ε, αυτή τη στιγμή έχουμε φτάσει σε μια πολύ καλύτερη κατάσταση και είναι πολύ περισσότερες οι χώρες, 12 ε, χώρες οι οποίες έχουν ε, διαδικασίες για μακροοικονομικά ελλείμματα τα δημοσιονομικά προγράμματα 10 χωρών ε, δεν ε, συμμορφούνται ε, με την φορολογική βάση. Τρία συμμορφούνται αλλά όχι πλήρως και δύο βρίσκονται σε κίνδυνο. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να ληφθούν επιπλέον μέτρα. Όχι βεβαίως να ξεκινήσουμε μια διαδικασία λόγω υπερβολικού ελλείμματος, αλλά εν πάση περιπτώσει ε, κάποιες συστάσεις έχουν γίνει. Επίσης έχει υπάρξει μία ε, αποκλιμάκωση της, ε, και μία επιβράδυνση μάλλον της οικονομίας και αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει έναν τρόπο να προχωρήσει κανείς αλλά πιστεύουμε ότι αυτός δεν είναι και ο καλύτερος, σωστό, ο καλύτερος τρόπος. Ο καλύτερος τρόπος είναι μέσα από μεταρρυθμίσεις οι οποίες δίνουν την δυνατότητα να αντιμετωπιστούν και άλλα προβλήματα όπως το δημογραφικό δημογραφικό, η γύρανση του πληθυσμού, ε, ε, κλιματικά κτλ. Η Κομισιόν έχει δημιουργήσει και ε, μία ολόκληρη υπηρεσία υποστήριξης καθώς επίσης και ένα πρόγραμμα το οποίο υποστηρίζει 500 μεταρρυθμιστικά προγράμματα σε όλες τις χώρες. Και στην επόμενη περίοδο, 21 με 27, προτείνουμε και ένα νέο υποστηρικτικό πρόγραμμα της τάξης των 25 δις ευρώ. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, ε, το εξάμεινο ε, έχει επιτυχία γιατί ακριβώς ε, βασίζεται στα τρία στοιχεία τα οποία ανέφερα προηγουμένως. Και με τον τρόπο αυτό έχει, έχει βοηθήσει τη διαδικασία του εξαμήνου στη μείωση των μακροοικονομικών ελλείψεων. Μας έχει δείξει ότι μπορεί να λειτουργήσει ε, αυτή τη στιγμή η ευρωπαϊκή οικονομία ε, βρίσκεται σε πορεία ανάπτυξης με θετικά στοιχεία για έβδομη ε, συνεχή χρονιά, ενώ ταυτοχρόνως διαπιστώνουμε επιβράδυνση στις αναδυόμενες οικονομίες συμπεριλαμβανομένες και της Κίνας. Σε αυτό θα μπορεί κανείς βεβαίως να προσθέσει και το άγνωστο στοιχείο του Brexit. Άρα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Η υλοποίηση όμως δεν εξαρτάται μονάχα από το εξάμεινο, αλλά εξαρτάται και από την κάθε μία χώρα ξεχωριστά και οπωσδήποτε εξαρτάται από τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείτε εσείς στις χώρες σας τη θητεία σας και οι κυβερνήσεις σας, τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούν ε, τις αξιολογίες του εξαμήνου. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Ντομπρόφσκης. Επιτρέψτε μου τώρα να σας παρουσιάσω τον επόμενο μας ομιλητή. Πρόκειται για την κυρία Μαριάν Τάισεν, αρμόδια επίτροπο για το χαπαρτοφυλάκιο της απασχόλησης των κοινωνικών υποθέσεων των ε, επαγγελματικών και εργασιακών δεξιοτήτων και κινητικότητας. Έχετε το λόγο κυρία Επίτροπε, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Καλησπέρα σας αγαπητοί συνάδελφοι. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε που μου δίνετε το λόγο. Έχω υπάρξει ευρωβουλευτή για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα και γι' αυτό πρέπει να σας πω ότι νιώθω σαν στο σπίτι μου εδώ, σε αυτή την αίθουσα. Καλωσορίζω ιδιαίτερο θερμά τους εκπροσώπους των Εθνικών Κοινοβουλίων, και τους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής καθώς και τους εκπροσώπους της Επιτροπής των Περιφερειών. Πολλοί είστε βετεράνοι του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και για κάποιους από εσά αυτό μπορεί να ηχεί ως κάτι το νέο και καινούριο, όμως για όλους εσάς είμαι πεπισμένη ότι το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο είναι εξαιρετικά σημαντικό, διότι στόχος του είναι να συντονίσει τις οικονομικές και κοινωνικές πολιτικές σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το εξάμεινο μας βοηθάει να μάθει ο ένας από τα λάθη του άλλου, να μάθει ο ένας από τις γνώσεις του άλλου, να βρούμε λύσεις και να ανοίξουμε ένα κοινό δρόμο στον οποίο θα πορευτούμε προς τα εμπρός. Είναι ένα πλαίσιο για την ανάλυση, για τον συντονισμό και τελικά για τις συστάσεις πολιτικής. Κάτι το οποίο μεταφράζεται σε μεταρρυθμίσεις οι οποίες θα είναι προσαρμοσμένες στις εκάστοτε εθνικές συντάσεις συνθήκες. Ω εργαλείο οικονομική διακυβέρνηση, το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο ήταν επιτυχία. Μα βοήθησε να φέρουμε σε πέρα μεγάλε μεταρρυθμίσεις, να φέρουμε την ανάκαμψη τη οικονομία και να καταστήσουμε τι οικονομίε μα πιο ανθεκτικέ. Τώρα όλε οι οικονομίε τη Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν ρυθμό ανάπτυξη και 240 εκατομμύρια Ευρωπαίοι εργάζονται, περισσότεροι από ό,τι οποτεδήποτε πριν στο παρελθόν. Ωστόσο, η Ευρώπη δεν σημαίνει μόνο τράπεζες και επιχειρήσεις. Ευρώπη σημαίνει κυρίως και πρώτα απ' όλα άνθρωποι. Άνθρωποι και γι' αυτό αυτή η Επιτροπή έχει διασφαλίσει ότι το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο δεν έχει μόνο να κάνει με την οικονομική και χρηματοπιστωτική μεταρρύθμιση, αλλά και με την κοινωνική μεταρρύθμιση. Και αυτό κατέστη ακόμα πιο σαφές, διότι συνδέθηκε το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο με τον Ευρωπαϊκό Πυλώνα Κοινωνικών ή Εργασιακών Δικαιωμάτων. Αυτός ο πυλώνας είναι ένα πλαίσιο 20 αρχών και δικαιωμάτων που ε, στρέφονται γύρω από τρεις βασικούς άξονες. Ίσες ευκαιρίες και ίση πρόσβαση στην αγορά εργασίας για να μπορούν όλοι να συμβάλλουν στην κοινωνία μέσω της δουλειάς τους, να μπορούν όλοι να έχουν τις δεξιότητες και τις ευκαιρίες να επιτύχουν. Δεύτερος άξονας είναι οι δίκαιες ηθίκες εργασίας, διότι το να έχει κανείς μια δουλειά δεν αρκεί πάντοτε θα πρέπει οι συνθήκες απασχόλησης να είναι δίκαιες και αυτό σημαίνει υψηλό επίπεδο ε, προστασίας ε, και ασφάλειας και σωστή ισορροπία μεταξύ οικογενειακής και προσωπικής ζωής από τη μία και επαγγελματική ζωής από την άλλη. Και τρίτος άξονας είναι η πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας, στις ε, υπηρεσίες προστασίας και βοήθειας για θέματα οικογένειας και τέκνων και ε, πρόσβαση σε ένα δίκαιο συνταξιδοτικό σύστημα. Σε κάθε περίπτωση μετά την οικονομική κρίση έχουμε επιταχύνει τις, ε, το ρυθμό μας για να μπορούν οι άνθρωποι να προσαρμοστούν στις επικείμενες αλλαγές που θα έρθουν στον ε, κόσμο της εργασίας. Αγαπητοί συνάδελφοι, αυτός ο πυλώνας εργασιακών δικαιωμάτων είναι κάτι το πολύ σημαντικό και τα τρία θεσμικά όργανα από κοινού προκήρυξαν τον Ευρωπαϊκό Πυλώνα στο, στη Σύνοδο του ε, Γκέτεμπουργκ το Νοέμβριο του 2017. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή άρχισε να χτίζει τον πυλώνα, να τον υψώνει σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και σε συνεργασία με το Συμβούλιο εκ μέρους 28 κρατών μελών. Ο πυλώνας αυτός συνοδεύτηκε από ένα νέο βαθμολόγιο, scoreboard, το οποίο πέρσι ενσωματώθηκε στο Ευρωπαϊκό Εξάμεινο και αυτό Μα δίνει μια άμεση επισκόπηση των κοινωνικών και εργασιακών μεταρρυθμίσεων που λαμβάνουν χώρα στα κράτη-μέλη. Φέτος λοιπόν διαπιστώσαμε πολύ σαφείς βελτιώσεις σε όλους τους βασικούς δείκτες κοινωνικής προόδου για την απασχόληση, για το ε, εισόδημα των οικοκυριών, για το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των δύο φύλων. Έχουν βελτιωθεί όλοι αυτοί οι δείκτες παντού. Το βαθμολόγιο μας δείχνει και τι προκλήσει που περιμένουν και που πρέπει να αντιμετωπίσουμε στα κράτη-μέλη που έχουν απομείνει έχουμε τις νέες ε, εκθέσεις αναχώρα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα τις δημοσιεύσουμε την επόμενη εβδομάδα και θα δείτε μεγαλύτερη προσοχή στις επενδύσεις στους τομείς προτεραιότητας για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτοί θα πρέπει να εμπνεύσουν και τον προγραμματισμό των Ταμείων Συνοχής ε, για το νέο επόμενο πολιετές δημοσιονομικό προγραμματικό πλαίσιο. Όλοι μοιραζόμαστε την ευθύνη, αγαπητοί συνάδελφοι. Έχουμε κοινή ευθύνη για μεταρρυθμίσεις με τον πυλώνα των εργασιακών δικαιωμάτων να είναι η πηξίδα μας, ο μπούσουλάς μας, το ευρωπαϊκό εξάμεινο και τα ευρωπαϊκά κονδύλια να είναι τα εργαλεία πλοήγησής μας, ανάλογα με τις ε, αρμοδιότητες του καθενός, της Επιτροπής, του Κοινοβουλίου και των κρατομελών και βεβαίως και των περιφερειών. Πλήρη στήριξη των κοινωνικών εταίρων και πλήρη στήριξη της οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών μας χρειάζεται. Ας εργαστούμε όλοι μαζί για να ε, έχει επιτυχία το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο, διότι μόνο μαζί από κοινού μπορούμε να διενεργήσουμε τις μεταρρυθμίσεις που χρειάζεται η Ευρώπη και τα κράτη-μέλη. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Η Πρόεδρος, και εγώ σας ευχαριστώ κυρία Επίτροπε. Επόμενος ομιλητής είναι ο κύριος Στίβεν Γκέραλντ που θα μιλήσει εξ ονόματος του κυρίου Τόμ Βαντεν ο οποίος ε, δυστυχώς δεν κατάφερε να ε, παραστεί. Σας δίνω το λόγο λοιπόν. Παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Επίτροποι, συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι. Προσωπώ το καλό μου φίλο, Τόμ Φαντενκέντελάρε, ο οποίος ασθενεί περαστικά Τόμ. Και έχει προετοιμάσει το, την ομιλία του στα αγγλικά και εγώ δεν μπήκα στον κόπο να τη μεταφράσω στη μητρική μου και θα το διαβάσω στα αγγλικά. Ως ε, εισηγητής της Επιτροπής ΕΚΟΝ για το Οικονομικό Εξάμεινο του 2019 θα ήθελε ο Τόμ να αναφέρει τις προτεραιότητες του. Ε, και ζητεί συγγνώμη για την αποσία του, αλλά ρώτησε το Σαββατοκύριακο και θα σας αναγνώσω εγώ τα σχόλιά του. Κυρίες και κύριοι, η συζήτηση που ασχολείται με το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο τίνει να είναι εξόχως πολιτική. Γι' αυτό είναι σημαντικό ε, να αφιερώσουμε χρόνο στις συζητήσεις αυτές και να ανταλλάξουμε τις κοινέ μας απόψεις μαζί με τα Εθνικά Κοινοβούλια. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το ίδιο, ο κύριος Λάρε, αυτό τον καιρό ολοκληρώνει την έκθεσή του. Ε, σε συνεργασία με διάφορες πολιτικές ομάδες και την άλλη εβδομάδα θα ψηφιστεί στην Επιτροπή ΕΚΟΝ και αρχές Μαρτίου θα συζητηθεί στην Ολομέλεια. Έχει έρθει η ώρα λοιπόν να μπούμε στις ίδιες προτεραιότητες. Η ετήσια μελέτη για την οικονομική ανάπτυξη Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχει θέσει προτεραιότητες και ο Επίτροπος Ντομπρόψης προηγουμένως αναφέρθηκε σε αυτές. Ε, υπάρχει μια πολιτική ε, καθοδήγηση γύρω από τρεις άξονες. Πρώτον, ε, δημοσιονομική εξυγίανση, δεύτερον, επενδύσεις και τρίτον, διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Δική μας δουλειά τώρα είναι να αναλύσουμε αυτό το τρίγωνο για να να έχουμε πιο μακροπρόθεσμες προτεραιότητες και να πούμε στο Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι ε, θεωρούμε σημαντικό και ποια είναι τα απαραίτητα βήματα πολιτικής που πρέπει να κάνουν. Ο Τόμ λοιπόν τονίζει μια πολύ μεγάλη πρόκληση. Η μακροπρόθεσμη προτεραιότητα είναι ο γυράσκων πληθυσμό. Και το σχέδιο έκθεσης του για το 2019, ο κύριος ε, Βαντανκέντελάρε θέλει ακριβώς να ασχοληθεί με αυτό το στοιχείο της γύρανσης του πληθυσμού και συγκεκριμένα τι αντίκτυπο θα έχει στα ασφαλιστικά συστήματα και στο κράτος πρόνοιας μας. Η δημογραφική αλλαγή είναι ένα ζήτημα αποφασιστικό εδώ και καιρό. Και δεν ε, συναντάει πάντα αυτό το πρόβλημα την νομοθεσία και την αντιμετώπιση στις πολιτικές. Θέλουμε λοιπόν να κληροδοτήσουμε ασφαλιστικά ταμεία και συστήματα στα παιδιά μας ή όχι. Αναφέρεται σε αυτό το θέμα το σχέδιο έκθεσης ε, και στην ετήσια έκθεση για την ανάπτυξη. Κάνει λόγο και για τις επενδύσεις και για τις διαρθωτικέ μεταρρυθμίσεις. Ε, τι συμβαίνει λοιπόν στις κοινωνίες μας που γυράσκουν γύρες του πληθυσμού είναι από τις σημαντικότερες δημογραφικές εξελίξεις και προκλήσεις του 21ου αιώνα και αφορά σχεδόν όλες τις χώρες του κόσμου. Αυξάνεται το προσδόκιμο ε, ζωής που βεβαίως αυτό σημαίνει ότι έχουμε περισσότερη ανάπτυξη και καλύτερα συστήματα υγείας. Αλλά έχουμε και προβλήματα, τα εξή δύο. Καθώς γυράσκει ο πληθυσμός, το κόστος για τις ε, συντάξεις, για την υγεία και για την ε, φροντίδα των ηλικιωμένων αυξάνεται. και είναι υψηλό ποσοστό του ΟΕΠ και αναμένεται να αυξηθεί ακόμα περισσότερο τις επόμενες δεκαετίες, διακυβεύοντας έτσι τη βιωσιμότητα των δημοσίων οικονομικών. Δεύτερον, δεν σημαίνει απλώς ότι αυξάνεται το κόστος, αλλά ότι μειώνεται και ο ρυθμός των εργαζομένων που βρίσκονται σε παραγωγική ε, ηλικία για να πληρώνουν τις συντάξεις. Πώς μπορούμε εμείς να προετοιμαστούμε για αυτές τις ε, προκλήσεις σύμφωνα με τον ΤΟΜ θα πρέπει να πιέσουμε τα κράτη-μέλη να ε, δημιουργήσουν πρώτα δημοσιονομικά μαξιλαράκια, κάποια αποθεματικά, στη συνέχεια να κάνουν ε, μεταρρυθμίσεις και τρίτον επενδύσεις ε, στραμμένες προς το μέλλον. Τι είναι αυτά τα δημοσιονομικά μαξιλαράκια. Θα πρέπει να έχουμε απόθεμα για να αντιμετωπίσουμε το την αύξηση των δαπανών που προέρχονται από τη γύρανση του πληθυσμού. Ιδιαίτερα σε καλούς οικονομικούς καιρούς χρειάζονται περισσότερες προσπάθειες. Αλλιώς θα κληρονομήσει η επόμενη γενιά το κόστος που θα είναι και αυξημένο. Το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης δεν είναι μόνο ποσοστά, είναι τα θεμέλια τα ίδια της νομισματικής μας ένωσης. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, οι κανόνες να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη αλλά και να εφαρμόζονται από όλα τα κρατη Δεύτερον, διαρθωτικές μεταρρυθμίσεις. Είναι σημαντικό να γίνουν αυτές ε, για να μειωθεί το κόστος ε, της γύρασης του πληθυσμού και να κινητοποιείται όσο γίνεται περισσότερο ο ενεργός πληθυσμός που μειώνεται έτσι κι αλλιώς. Ψηφιοποίηση, παγκοσμιοποίηση και τεχνολογικές αλλαγές ραγδαία μεταβάλλουν την αγορά εργασίας μας. Και αυτά επηρεάζουν τη φύση των εργασιών, των καθηκόντων ε, και των δεξιοτήτων και ικανοτήτων που απαιτούνται. Γι' αυτό χρειάζεται πιο μεγάλη ευελιξία στην αγορά και εργαζόμενοι που μπορούν να απασχολούνται σε διάφορες δουλειές. Επενδύσεις στο μέλλον. Η δικαιοσύνη μεταξύ των γενεών σημαίνει ότι θα πρέπει να εξασφαλίσουμε παραγωγικότητα και για το μέλλον για να είναι βιώσιμη η οικονομική ανάπτυξη και ε, να έχουμε παραγωγικές επενδύσεις στραμμένες στο μέλλον και οι δημόσιες και οι ιδιωτικές σε σχολεία, παιδεία, έρευνα, ανάπτυξη, έργα υποδομών αλλά επίσης και πιο σημαντικό ακόμα στην καινοτομία και την ψηφιοποίηση. Για να συνοψίσω, το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο θα μπει προσεχώς στις φάσεις της, ε, των συστάσεων αναχώρα. Θα κάνει πρώτα ανάλυση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μέχρι τα τέλη του μηνός θα την παρουσιάσει και στη συνέχεια θα καταθέσει τις συστάσεις αναχώρα ε, στις 29 Μαΐου. δεν είναι πολύ ενθαρρυντικά τα στοιχεία ως προς την εφαρμογή των συστάσεων αναχώρα. Βεβαίω θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι είναι συστάσει και όχι υποχρεώσεις δεσμευτικές για να γίνεται καλύτερη εφαρμογή και χρειάζεται πολιτική υποστήριξη σε όλα τα επίπεδα. Είναι αποφασιστική σημασία και έχουν κρίσιμο ρόλο εδώ να διαδραματίσουν τα εθνικά κοινοβούλια. Και έκφραση αυτού ακριβώ είναι τούτη εδώ η κοινοβουλευτική εβδομάδα. Και ε, περιμένω να ακούσω τι απόψει για το πώ θα προχωρήσουμε. Αυτά λέει ο Τόμ και ζητώ συγγνώμη που μακρηγόρησε. Ευχαριστώ. Thank you. Εγώ σας ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος. Τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στην επόμενη ομιλήτρια, είναι η κυρία Αγνιέσκα Κοσλόξα Ραγεύιτς, μέλος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβούλιο. Του Κοινοβουλίου, συγγνώμη. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Επίτροποι, αγαπητά μέλη του των Κοινοβουλίου, θα ήθελα να μιλήσω στα πολωνικά, γι' αυτό βάλτε όλοι τα ακουστικά σας. English is on the second canal. Szanowni Państwo, tegoroczny semestr europejski... Κυρίες και κύριοι, αυτό το ευρωπαϊκό εξάμεινο μας φέρνει ε, πολύ καλά νέα όπως μας τα παρουσίασαν άλλωστε και οι εκπρόσωποι της Επιτροπής. Ωστόσο φέρνει και πολλές προκλήσεις οι οποίες απαιτούν προσπάθειες ε, διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η μόνη οικονομία του κόσμου που συνδυάζει την ευημερία με την προστασία των εργαζομένων και η ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης οφείλει να είναι ε, δίκαιη και φιλική προς το περιβάλλον, άρα και οικολογική. Θα πρέπει επομένως να γίνει προσπάθεια έτσι ώστε να συνδυαστούν πολλά ε, ε, στοιχεία. Στο ε, εξάμεινο αναγνωρίζονται βεβαίως θετικά στοιχεία όσον αφορά την αγορά εργασίας, ας πούμε, μείωση της ανεργίας. Υπάρχουν καλά αποτελέσματα επίσης όσον αφορά την ευρωπαϊκή οικονομία. Ωστόσο, αυτά τα καλά αποτελέσματα δεν αφορούν όλους τους πολίτες της Ευρώπης. Εξακολουθούν να υπάρχουν διαφορές σε επίπεδο περιφερειών αλλά και σε επίπεδο χωρών. Είναι πολλά εκατομμύρια οι άνθρωποι αυτοί, οι πολίτες αυτοί, οι οποίοι κινδυνεύουν με κοινωνικό αποκλεισμό. Επίσης, 6 εκατομμύρια ε, νέοι αντιμετωπίζουν νεανική ανεργία. Από την άλλη πλευρά διαπιστώνουμε ότι ε, αυξάνει ε, και η διαφορά ε, το, της απασχόλησης ανάμεσα σε γυναίκες και άνδρες. Είναι πολλές ε, οι γυναίκες μιας κάποιας ηλικίας ε, οι οποίες αποφασίζουν να εγκαταλείψουν την ενεργό ας πούμε ζωή για να ασχοληθούν με την οικογένειά τους. Θα πρέπει οπωσδήποτε να θέσουμε με μεγάλη ρόμη και μετεπιτάσεως το θέμα της, ε, των, των ε, ε, γερόντων, το θέμα των ανθρώπων προχωρημένης ηλικίας και αυτών που θα τους προσέχουν. Επίσης, ε, το θέμα της ε, ε, εργασίας των οικιακών βοηθών. Πολύ συχνά δουλεύουν στην μαύρη εργασία. Όχι γιατί το θέλουν και γιατί είναι η επιλογή τους, αλλά σε πολλές περιπτώσεις και σε πολλές χώρες δεν προβλέπονται οι σωστές συνθήκες έτσι ώστε να μην δουλεύουν στην μαύρη αγορά ε, η οικιακή βοηθή. Ε, εξακολουθεί επίσης να υπάρχει διαφορά ανάμεσα στις γυναίκες και τους άνδρες και γι' αυτό λέμε ότι η απασχολησιμότητα των γυναικών μπορεί να αυξηθεί μονάχα και εφόσον δημιουργηθούν ε, οι δομές φύλαξης των παιδιών. Και επομένως εδώ έχουμε και ε, σχετικές ε, προτάσεις οι οποίες θα φτάσουν οπωσδήποτε ε, ακολουθώντας τη συνήθη πορεία και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα πρέπει να συνδυαστεί η επαγγελματική ζωή με την οικογενειακή ζωή. Η συμφιλίωση αυτή είναι πάρα πολύ σημαντική αν θέλουμε να μιλήσουμε για την αγορά εργασίας. Ένα άλλο κλειδί για την αγορά εργασίας είναι η εκπαίδευση. Γνωρίζουμε ότι 40% των εργοδοτών δεν καταφέρνουν να βρουν καταρτισμένο προσωπικό, ακριβώς όπως το θέλουν. Άρα υπάρχει μια διαφορά ανάμεσα από τις δεξιότητες τις οποίες μαθαίνουν ε, οι νέοι ε, και ε, τις δεξιότητες τις οποίες η αγορά εργασίας ζητά. Επίσης, 30% ε, των ε, ανθρώπων στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ε, γνωρίζουν, δεν έχουν ψηφιακές ικανότητες. 20% δεν έχουν καλές ικανότητες όσον αφορά την ανάγνωση, τον αλφαβητισμό γενικά. Ένα από τα πιο σημαντικά προγράμματα, σχέδια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Συμβουλίου αφορά ακριβώς την αγορά εργασίας και σχετίζεται ακριβέστατα με το θέμα που ανέφερα προηγουμένως, δηλαδή της προσαρμογής των δεξιοτήτων. Κύριο μέλημα είναι ε, η αύξηση των ε, soft, των υπείων ικανοτήτων. Θα πρέπει οπωσδήποτε επίσης να ε, δώσουμε μεγάλη σημασία στην διαβίου εκπαίδευση και την διαβίου κατάρτιση. Επίσης, η ψηφιακή μετάβαση είναι κάτι που πρέπει να προετοιμάσουμε προσεκτικά. Ε, επίσης, ε, να μην ε, λησμονούμε ότι και στο τομέα αυτό οι δεξιότητες των γυναικών υπολείπονται των δεξιότητων των ανδρών. Λίγες είναι οι γυναίκες που κάνουν, ας πούμε, e-banking. Είναι λίγες οι γυναίκες οι οποίες ασχολούνται με την τεχνολογία, με την πληροφορική, με τις επικοινωνίες. Ωστόσο, αυτά ακριβώς τα στοιχεία αποτελούν τη βάση για το μέλλον. Εμείς δεν θέλουμε το μέλλον να οικοδομηθεί μονάχα επί των ανδρών. Ε, θέλουμε και τις γυναίκες στη διαδικασία αυτή. Και ε, με την ε, οδηγία η οποία ο Σονούπο θα έρθει και στο Κοινοβούλιο για την αγορά εργασίας οπωσδήποτε θα καταφέρουμε να βελτιώσουμε την κατάσταση. Επίσης η κατάσταση θα βελτιωθεί εάν σπάσουμε και τα στερεότυπα και τότε ε, δεν θα είναι μονάχα κοινωνικό ε, το κέρδος, αλλά θα έχουμε και περισσότερες γυναίκες στην αγορά εργασίας και θα έχουμε και καλύτερη αντιστοίχηση των ε, ε, δεξιοτήτων που αναζητούν οι εργοδότες με αυτές που έχουν οι εργαζόμενοι και θα έχουμε μια πραγματικά ανοιχτή και ευημερούσα Ευρώπη. Ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ. Επόμενη ομιλήτρια η Μαρία Ντελμάρ Άγκουλο από το Ισπανικό Κοινοβούλιο. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα καταρχάς να σας ευχαριστήσω γιατί μου δίνετε την δυνατότητα να συμμετάσχω σε αυτή τη ε, συζήτηση για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο ως εργαλείο συντονισμούς. Είμαστε στο τέλος μιας ε, κοινοβουλευτικής θητείας με νέο ορίζοντα για τον προπολογισμό και με τους ε, στόχους στραμμεσμένους στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής για την Ευρώπη το 2020. Εννέα χρόνια μετά τη δημιουργία του το 2010, το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο έχει αποδείξει κάτι πολύ σημαντικό. Επιτρέπει στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να σχεδιάσουν τις προϋπολογιστικές τους προτάσεις από τη στιγμή που θα γνωρίζουν τις λεπτομέρειες για τις προτεραιότητες δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι δεν υπάρχουν κίνδυνοι αμφιβολιών που να του επηρεάζουν τις χώρες μέλη ή ενδυνάμει ανισορροπίας ανισορροπίες. Ε, τα πράγματα γίνονται καλύτερα, είναι πιο ξεκάθαρα και είναι πιο εύκολο να έχουμε μια σωστή οικονομική πολιτική και χρηματοπιστωτική πολιτική. Είναι περισσότερες οι εγγυήσει που προσφέρονται στους πολίτες. Έχουμε μεγαλύτερη εμπλοκή, αν όχι και συνενοχή μεταξύ ε, ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων με τους Ευρωπαίους πολίτες και την οργανωμένη κοινωνία των πολιτών. Όλοι αυτοί δηλαδή γίνονται σύμμαχοι και συντάσσονται στην ίδια, πίσω από τις ίδιες τάξεις, πίσω από τις ίδιες γραμμές. Το σημαντικό είναι οι στόχοι έτσι όπως έχουν τεθεί. Είναι αντικειμενικό λοιπόν να πει κανεί ότι έχουμε προχωρήσει σημαντικά στις τέσσερις γραμμές του προπολογισμού που είχαν τεθεί εξ αρχή. Την εξυγίανση των δημοσίων οικονομικών με έξι ποσοστιαίες μονάδες βελτίωση, και την εξυγίανση των καταστάσεων και έχουμε αποφύγει μακροοικονομικές ανισορροπίες, τις έχουμε διορθώσει, έχουμε ενθαρρύνει την επένδυση και έχουμε δώσει πρωταρχικό ρόλο στις διευθυντικές μεταρρυθμίσεις που δημιουργούν θέσεις απασχόλησης. Και ο πρόεδρος Γιούγκερ στην ομιλία του πρόσφατα το ανέφερε. Έχουμε 23 τρίμενα συνεχούς ανάπτυξης και δημιουργία 12 εκατομμυρίων θέσεων εργασίας. Όλα αυτά είναι πολύ εύγλωτα. Το, από το Δεκέμβριο του 2011 μέχρι τον Μάιο του 2018 μειώθηκε το έλλειμμα στην Ισπανία πάνω από 6 ποσοστιαίες μονάδες. Ε, ε, δημιουργήθηκαν 3,4 εκατομμύρια θέσεις εργασίας και είχαμε ρυθμό ανάπτυξης που άγγιζε το 3,1%. Όλα αυτά λοιπόν δείχνουν τις θετικές εξελίξεις και πόσο θετική ήταν η συμβολή και η συνεισφορά του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Δεν πρέπει βεβαίω να είμαστε αυτάρεσκοι και να ικανοποιούμαστε με, τα, με τη δουλειά μας μόνο. Προχωρώντας σε αυτόν τον δρόμο θα φτάσουμε τελικά στον επιθυμητό προορισμό, απλουστεύοντας τις διαδικασίες, βελτιώνοντας την επικοινωνία. Σε κάθε περίπτωση ήταν θετικός ο αντίκτυπος του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Από εκεί και πέρα, το εξάμεινο απέδειξε τη δύναμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία μπορεί να δώσει απαντήσεις. Η οικονομική κρίση ήταν πρόκληση πρώτη τάξη για την Ευρώπη και μάλιστα ε, τέθηκε σε κίνδυνο και το χειρό του ευρώ, του ενιαίου νομισματο. Η κρίση είχε ε, συντριπτικό αποτέλεσμα στην κατάσταση των δημοσίων οικονομικών των χωρών και είχε και συντριπτικό αποτέλεσμα στην πραγματική οικονομία, γιατί είχαμε καταστροφή, κατάργηση θέσεων εργασία. και όλα αυτά χρειαζόντουσαν πολύ έγκαιρη και ταχεία απάντηση από δική μα πλευρά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν πρόσφερε εργαλεία για να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση, μέτρα για να ενισχυθεί η ίδια κυβέρνηση εκεί όπου είχαν υπάρξει αδυναμίες λόγω της κρίσης και υπ' αυτή την έννοια το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο αποδείχθηκε ως ένα εργαλείο πανίσχυρο, πολύ χρήσιμο για να δείξει στους πάντες ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σε θέση να κομίσει απαντήσεις. Τέλος, θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντική η δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η, η προσήλωσή της στη σταθερότητα, η ενίσχυση των συναγερμών, των προεδοποιήσεων, των προεδοποιητικών σημάτων. Όλα αυτά έχουν να κάνουν με την υπευθυνότητα, με τη λογοδοσία κατά, την, ε, ε, κατά το σχεδιασμό των προϋπολογισμών και έχουν να κάνουν με τη σταθερότητα περί των οικονομικών. Όλα αυτά αποτελούν εγγύηση για τον πολίτη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση με τις οικονομικές αξίες, με τη σταθερότητα, με ισορροπημένα δημόσια οικονομικά, πορεύεται με επιτυχία προς τα εμπρό και αυτά είναι οι βασικές εγγυήσεις για το κράτος πρόνοιας. Γιατί έτσι έχουμε αύξηση της κατανάλωσης, αύξηση των επενδύσεων και άρα έχουμε δέσμευση για το ότι η σταθερότητα θα φέρει θετικά ωφέλη και στην ανάπτυξη και στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Και ε, από εκεί και πέρα. Υπάρχει δέσμευση εναντί των δράσεων των κρατών των μελών, τα οποία κράτη-μέλη είναι σταθερά προσιλωμένα στις μεταρρυθμίσεις. Πάντοτε έχουμε απαιτήσει και τις συνδέουμε με τη στήριξη προς το κράτος και στηρίζουμε το κράτος στο βαθμό που τηρεί τις απαιτήσει που περιμένει κανείς από αυτό. Αυτό το δίδυμο λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό ε, κατά την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων και θέλω να αναφερθώ στην υπηρεσία στήριξης διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς τα κράτη-μέλη. Είναι πολύ υψηλή η ζήτηση για τις ε, υπηρεσίες αυτού του τμήματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και πολύ σημαντικό το έργο που παράγει. Έχουμε επίση και δράση για τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Γίνονται προσπάθειες και μεταρρυθμίσεις σε μία κρατός μέλο, και αυτό έχει πολλαπλασιαστικό όφελο στα άλλα κράτη-μέλη γιατί έτσι μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να σχεδιάζει με μεγαλύτερη συνέπεια και συνοχή στον τρόπο σκέψη τη. Τέλο. κυρίες και κύριοι, θα πρέπει οι πολίτες να καταλάβουν πολύ καλά ότι η Ευρώπη είναι η εγγύηση για την απάντηση στα προβλήματα των πολιτών και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα γίνει πανίσχυρη όταν αποδείξει πλέον την δυνατότητά της να συνεργάζεται και να προσφέρει λύσεις. Και άρα έχουμε πολύ χρήσιμα εργαλεία που πρέπει να τα τονίσουμε, να τα φέρουμε στο προσκήνιο. Το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο είναι ένα τέτοιο εργαλείο και με τις τροποποίησεις και με τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις που θα κάνουμε αξίζει να συνεχίσουμε να το χρησιμοποιούμε αυτό το εργαλείο που μας ωφελεί τόσο πολύ. Σας ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Τελευταίος αλλά όχι λιγότερο σημαντικός, ο κύριος Τζον Λαχάρτ, μέλος της Ιρλανδικής Βουλής. Έχετε παρακαλώ το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την ευκαιρία που μας δίνετε να μιλήσουμε στην εναρκτήρια συνεδρίαση. Λέγομαι Ζων Λαχάρτ, αντιπρόεδρος της Επιτροπής ε, Δημοσιονομικού Ελέγχου της Ιρλανδικής Βουλής σε ό,τι αφορά το ευρωπαϊκό εξάμεινο και τι σημασία έχει για τον προπολογισμό, θα πρέπει να εξηγήσουμε ότι τα τελευταία χρόνια η Ιρλανδική Βουλή έκανε βήματα για να αναθεωρήσει τον τρόπο με τον οποίο εξτάζει τον προπολογισμό. Τμήμα αυτών ήταν η ε, ίδρυση γραφείου προπολογισμού στη Βουλή του 2017. Ως αποτέλεσμα τώρα οι Ιρλανδοί βουλευτές έχουν πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας ε, έρευνα και πραγματογνωμοσύνη και ελέγχουμε βασικά έγγραφα του προπολογισμού πολύ περισσότερο από ό,τι στο παρελθόν. Η Επιτροπή μας επίσης ιδρύθηκε ε, με τη μεταρρύθμιση αυτή για να συμμετέχει περισσότερο η Βουλή σε ολόκληρη τη δημοσιονομική διαδικασία. Η Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού συνεργάζεται με το Γραφείο Προπολογισμού της Βουλής για να ε, βελτιώνεται η ενημέρωση στους βουλευτές ως προς τον βιολογισμό και να γίνεται ο έλεγχος εκ των προτέρων, πολύ νωρίτερα από την κατάρτιση του προπολογισμού. Ακόμα είμαστε στα σπάργανα. Ε, επίσης, για να βάλουμε τα θεμέλια για να υπάρχει ουσιαστικός κοινοβουλευτικός δημοσιονομικός έλεγχος, η Επιτροπή μας άρχισε να ευθυγραμμίζεται με το χρονοδιάγραμμα του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και ε, σε συνεργασία με την Επιτροπή Οικονομικών βέβαια της Βουλής. Δηλαδή έχουμε τακτικές επαφές ε, ευρωπαϊκών ε, στελεχών κάθε χρόνο το Απρίλιο συζητούμε με τον Υπουργό Οικονομικό το πρόγραμμα σταθερότητας πριν υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και οι δύο επιτροπές επίσης συναντήθηκαν με τον Επίτροπο Ντομπρόφσκης και την Επιτροπή Προϋπολογισμών για να συζητήσουν το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2020-2027 και την αναθεώρηση του κοινοτικού προϋπολογισμού. Επίσης, τον Απρίλιο συναντηθήκαμε για να συζητήσουμε τις εκθέσεις και τις συστάσεις αναχώρα. Και τον άλλο μήνα ε, πρόκειται να συναντηθούμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, για να εκτάσουμε την έκθεση για την Ιρλανδία. Ανταλλάσσουμε απόψεις λοιπόν με τον Υπουργό Οικονομικό επίσης όταν παρουσιάζει το πρόγραμμα σταθερότητας και έχουμε μια μόνιμη αλληλεπίδραση με το αρμόδιο Οικονομικό Συμβούλιο της χώρας. Και η Επιτροπή ε, προπολογισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ο κύριος Ντομπρόφσκης ε, συμμετείχαν στο παρελθόν ε, στις εργασίες μας και θέλω να τους ευχαριστήσω. Και προσβλέπουμε στη μελλοντική συνεργασία μας. Σε ό,τι αφορά στην εθνική διαδικασία του προπολογισμού, του Ευρωπαϊκού Εξάμεινο αποτελεί ένα σημαντικό πλαίσιο για τη συνολική κατάρτιση του εθνικού προπολογισμού όλο και περισσότερο θέλει να συμμετέχει το Κοινοβούλιο στο Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Α πούμε, η ενημέρωση του προγραμμάτου σταθερότητα θα συζητηθεί στο Κοινοβούλιο και στη δική μα Επιτροπή. Ε, συνεργαζόμαστε με το ε, Συμβουλευτικό Οικονομικό Συμβούλιο και βλέπουμε και πώς ε, επηρεάζουν ε, τον προπολογισμό της χώρας όλες οι ευρωπαϊκές διαδικασίες. Θα πρέπει να εστιάσουμε περισσότερο στην ποιότητα των πληροφοριών για τον προπολογισμό σε έγγραφα πριν ε, την κατάρτιση του προπολογισμού και συζητούμε εγκαίρως και εκ των προτέρων κάθε χρόνο το θέρος. Γι' αυτό λέγεται και θερινό πρόγραμμα. Υπάρχει χώρος βέβαια πάντα για βελτίωση και για μεταρρυθμίσεις και συνεργάζομαι με τους συναδέλφους στην Επιτροπή μας και έχουμε μάθει περισσότερα για την προσήλωση της Ιρλανδίας στο Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Αυτό είχε και θετική ε, απήχηση ε, στον προπολογισμό της χώρας. Ενθαρρύνθηκε και η διαφάνεια και η κοινοβουλευτική διαδικασία και ο διάλογος στο Κοινοβούλιο. Πώς μπορεί να βελτιωθεί τώρα το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Ε, το χρονοδιάγραμμα καμιά φορά δεν επιτρέπει πλήρη συμμετοχή του Κοινοβουλίου στο προσχέδιο προπολογισμών, α πούμε, πέρυσι δεν είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, γιατί είχε ε, προβλεφθεί συζήτηση την 9η Οκτωβρίου του 2018, που είναι η μέρα του προπολογισμού στην Ιρλανδία. Χρειάζεται νωρίτερα να προγραμματίζεται αυτή η διαδικασία, συνάδοντας με οικονομικούς κύκλους. Αυτό θα μπορούσε να το εξτάσει το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Επίσης, μπορεί να χρειαστεί μεγαλύτερη ευελιξία στην εφαρμογή των δημοσιονομικών κανόνων, ε, ιδιαίτερα σε ό,τι ε, αφορά ε, ένα μέτωπο για την αντιμετώπιση ε, των δυσμενέστερων ε, εποχών. Στι συστάσει αναχώρα και στην έκθεση αναχώρα επίσης είναι σημαντικό να συμμετέχουν τα κοινοβούλια. Έχουμε αρχίσει να συζητούμε αυτά τα στοιχεία και θα εξακολουθήσουμε να συμμετέχουμε στη συζήτηση στο Κοινοβούλιο της Ελλάδας. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, και εγώ σας ευχαριστώ και θα ήθελα τώρα να ευχαριστήσω όλους τους ομιλητές μας, τους διακεκριμένους ε, προσκεκλημένους για τις απόψεις τους και τις ε, μεστές ε, παρουσιάσεις και θα δώσω το λόγο και πάλι στο συμπρόεδρο, τον κύριο Ρομπέρτο Γκουαλτιέρη. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Thank you very much. Σας ευχαριστώ πολύ. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν τώρα τη συζήτηση. Ο κύριος Φέιλερ από την Γερμανία και το ΕΛΚ είναι ο πρώτος που θα πάρει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο εισήχθη ως μηχανισμός προειδοποίησης ε, στις εποχές ε, της κρίσης. Μάθαμε ότι είναι επιτυχία ακόμα και συμφωνώ γιατί μετεξελίχθηκε υπήρξε συνέχεια, ανανέωση και δουλειά επί του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Πού θα βρισκόμαστε εάν δεν υπήρχε το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο ε, και αν δεν είχε εφαρμοστεί 30-40% αλλά περισσότερο, όπως και οι συστάσεις χώρα. θα είχαμε προχωρήσει ακόμα περισσότερο. Ε, Παρ' όλα αυτά, η οικονομική ανάπτυξη δεν φτάνει σε όλους τους Ευρωπαίους πολίτες ε, με τον ίδιο τρόπο και στον ίδιο βαθμό. Στη Γερμανία, ας πούμε, ανεβήκαμε πολύ ψηλά με την οικονομική μας ανάπτυξη και σιγά σιγά αρχίζει η ύφεση, ε, γιατί έχουμε τεράστια έλλειψη εργαζομένων. Αλλού υπάρχει μεγάλη ανεργία το ακούσαμε ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την ανεργία των νέων. Έχουμε μεγάλες προκλήσεις, ε, διαρκώς αυξανόμενες και τα κράτη-μέλη ε, δεν θα πρέπει να χαλαρώσουν στις προσπάθειες για μεταρρυθμίσεις. Χρειάζονται στοχευμένες επενδύσεις, μείωση του χρέους και φυσικά ε, αυτό το buffer, το μαξιλαράκι στον προϋπολογισμό. Σημαντικά στοιχεία για τη σταθερότητα. Θα ήθελα να κάνω μία πρόταση εδώ. Τα κονδύλια της συνοχής θα πρέπει να συνδέονται πιο στενά με το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο και με τις μεταρρυθμίσεις. Ε, οι μεταρρυθμίσεις διαρθρωτικές θα πρέπει να προσανατολίζονται στις τάσεις αναχώρα για να δημιουργηθεί ένα υγιές τοπίο και περιβάλλον για τις επενδύσεις. Ευχαριστώ πολύ. Thank you very ευχαριστώ. Ο κύριος Ανισλάβεκ από την Πολωνία, ECR. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, κανείς από μας δεν αμφιβάλλει για τα θετικά στοιχεία που μπορεί να έχει στην οικονομία της Ένωσης ε, το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Οχτώ χρόνια λειτουργίας αυτού του μηχανισμού νομίζω ότι αρκούν έτσι ώστε να έχουμε μια σε βάθος ε, συζήτηση για αυτό το εξάμεινο ε, όσον αφορά τα νέα σενάρια μετά από το 2020. Θα πρέπει να δούμε δηλαδή εάν η παρούσα πρακτική του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου μπορούν να ευθυγραμμιστούν και να ανταπεξέλθουν ε, στις νέες προκλήσεις που θα αντιμετωπίσουν τα κράτη-μέλη και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το σύστημα συντονισμού των οικονομικών πολιτικών είναι πολύ καλό εάν εάν υπάρχει ένα αποτελεσματικό ε, σύστημα ε, που θα, μπορούσαν, ε, που θα μπορούσε να βοηθήσει τις χώρες αυτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίες αντιμετωπίζουν μεγάλες απώλειες τότε αυτό θα ήταν πάρα πολύ καλό Βεβαίως εδώ μιλάμε για θέματα δύσκολα και ευαίσθητα και ίσως δεν είναι και ο δικός μας λόγος σαν ε, ρόλος ως εθνικοί βουλευτές να ασχοληθούμε με τα θέματα αυτά. Μερικές φορές ε, είναι γεγονός ότι απλά μαθαίνουμε κάποιες πληροφορίες από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή την ε, Κομισιόν, ενώ πιστεύω ότι θα πρέπει να παίξουμε ένα πιο ενεργητικό ρόλο όσον αφορά την σωστή οικονομική διακυβέρνηση, διακυβέρνηση, την governance και οπωσδήποτε θα πρέπει να προσπαθήσουμε να βρούμε κοινέ λύσεις για αυτά τα προβλήματα που είναι κλειδιά για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ίσως κάθε φορά που συναντιόμαστε θα πρέπει να συμπεριλαμβάνουμε και μία στιγμή ε, συγκεκριμένης ψηφοφορίας, επίσημης ψηφοφορίας, ε, για να δούμε πόσοι συμφωνούν με κάποιες προτάσεις, έστω και αν αυτές δεν είναι υποχρεωτικές. Υπενθυμίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συχνά επιλέγει την συναπόφαση για τα πιο ευαίσθητα θέματα και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι η πρώτη η οποία ε, θέλει να προωθήσει την βαθμιαία πλειοψηφική ψήφο έναντι της ομοφωνίας σε μία σειρά θεμάτων. Έχουμε και τον ε, Επίτροπο Μοσχοβησί, ο οποίος λέει ότι είχε έννοια η ομοφωνία την ε, δεκαετία του 50, αλλά ήταν και λίγες οι χώρες, ενώ τώρα δεν είναι πλέον επίκαιρη αυτή η διαδικασία, είναι μάλλον αναχρονιστική. Θα πρέπει να προετοιμάσουμε και να προετοιμαστούμε μάλλον κατά την έννοια αυτή και προς αυτήν την κατεύθυνση. Και βεβαίως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Ρουμανική Προεδρία θα μπορούσε να οργανώσει μια ομάδα εργασίας έτσι ώστε να αξιολογηθούν σωστά τα όσα έγιναν τα τελευταία 8 χρόνια. Ευχαριστώ. Σα... Σας ευχαριστώ. Καλωσορίζω πολύ αυτό που λέτε για την ειδική πλειοψηφία στη ψηφοφορία. Για να γίνει κάτι τέτοιο σε αυτή τη συνεδρίαση θα πρέπει να γίνει στάθμιση μεταξύ των χωρών. Πολύ δύσκολο το εγχείρημα, αλλά είναι ενδιαφέρουσε οι προτάσει. Ο κύριο Παπαδημούλη είναι ο επόμενο ομιλητή από την ΚΟΕ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ξεκινήσω με κάποια νέα από τη χώρα μου την Ελλάδα. Οι τελευταίες προβλέψεις της Κομισιόν προβλέπουν ρυθμό ανάπτυξης στην Ελλάδα για το 2019 2,4%. Μετά από πολλά χρόνια κρίσης η χώρα μου έχει μπει σε ρυθμούς ανάπτυξης της οικονομίας της ψηλότερες από το μέσο όρο της Ευρωζώνης και οι ίδιοι ρυθμοί προβλέπονται για τα έτη 2020 και 2021. Και έχουμε και μια αύξηση των επενδύσεων και μια σημαντική μείωση της ανεργίας που παραμένει όμως ακόμη υψηλή. Θα ήθελα να πω όμως ότι στις ίδιες προβλέψεις της Κομισιόν προβλέπεται μια επιβράδυση της οικονομίας για το σύνολο της Ευρωζώνης σε σχέση με τις προηγούμενες προβλέψεις. Επιβράδυση για τη γερμανική οικονομία, για την γαλλική οικονομία, για την ιταλική οικονομία. Πράγμα που σημαίνει ότι πρέπει να κάνουμε περισσότερα και καλύτερα ως χώρες της Ευρωζώνης για να αντιμετωπίσουμε την πιθανή κρίση που έρχεται εξαιτίας και της διεθνούς αβεβαιότητας και των εμπορικών πολέμων που είναι επιθύρες ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα για παράδειγμα. Και από αυτή την ε, σκοπιά θα ήθελα να επισημάνω ότι έχει ιδιαίτερη σημασία η Ρουμανική Προεδρία και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα Εθνικά Κοινοβούλια να πιέσουμε έτσι ώστε να ολοκληρωθούν επιτέλους οι διαπραγματεύσεις για το νέο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο για τα έτη 2021-2027. Στην Κομισιόν και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουμε ένα προσανατολισμό συγκεκριμένο, αλλά δυστυχώς υπάρχουν ορισμένα κράτη-μέλη στο Συμβούλιο, ορισμένες κυβερνήσεις, οι οποίες καθυστερούν και αναβάλουν. Και η καθυστέρηση κάνει ζημιά στην οικονομία. Το δεύτερο πράγμα που θέλω να επισημάνω είναι ότι επί τέσσερα χρόνια παρότι το Κοινοβούλιο και η Κομισιόν πιέζουν, δεν έχει ολοκληρωθεί η τραπεζική ενοποίηση. Γιατί δεν έχουν γίνει βήματα για την υλοποίηση του τρίτου πυλώνα τη τραπεζική ενοποίηση που αφορά το ευρωπαϊκό σύστημα εγγύησης καταθέσεων. Δυστυχώ υπάρχουν ορισμένε κυβερνήσει και ονομάζω συγκεκριμένα οι κυβερνήσει τη Ολλανδίας και τη Γερμανία που αρνούνται να ολοκληρωθεί η τραπεζική ενοποίηση. Το τρίτο θέμα που νομίζω ότι πρέπει να μας απασχολήσει είναι η φορολόγηση της ψηφιακής οικονομίας. Είναι αδιανόητο οι γίγαντες του ίντερνετ να μην πληρώνουν καθόλου φόρο, ενώ οι μισθωτοί, οι συνταξιούχοι, οι ελεύθεροι επαγγελματίε, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις πληρώνουν πάρα πολλούς φόρους. Και για να γίνει αυτό χρειάζεται μεγαλύτερη συνεργασία ευρωπαϊκή και φορολογική εναρμόνιση. Μόνο έτσι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε και τις μεγάλες ανισότητες που στα χρόνια αυτά μεγαλώνουν και ανάμεσα στους πλούσιους και τους φτωχούς και ανάμεσα στα πλουσιότερα κράτη-μέλη και στα φτωχότερα κράτη-μέλη και ειδικά για την πολιτική συνοχής. Θεωρώ αδιανόητο να περικόπτονται κονδύλια από την πολιτική συνοχής στο νέο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Εμβληματικές πολιτικές όπως η κοινή αγροτική πολιτική και η πολιτική συνοχής πρέπει να ενισχύονται και όχι να αποδυναμώνονται, γιατί η αποδυνάμωση αυτών των πολιτικών τους μόνους που τρέφει είναι τους ακροδεξιούς λαϊκιστές που θέλουν τη διάλυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας ευχαριστώ. Thank you. Ευχαριστούμε πολύ. Μαργαρίτα Μάρκε από την Πορτογαλία και την πολιτική ομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο έχει γίνει η πιο σημαντική άσκηση συντονισμού πολιτικών οικονομικών και κοινωνικών και εργασιακών. Έχει γίνει μέρος της καθημερινότητάς μας, της καθημερινής ένομης τάξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση για όλα τα κρατημέλη που είναι μέλη αυτής. Πολύ συχνά γίνεται λόγος για την ανάγκη να προσεγγίσουμε την Ευρώπη των πολιτών, να, να κάνουμε την Ευρώπη να πλησιάσει τους πολίτες και να γίνει πιο δημοκρατική. Είναι πολύ σημαντικό να γίνεται αυτή η συζήτηση τη στιγμή που γίνεται λόγος και εξετάζονται συγκεκριμένες πολιτικές. Ερωτώ λοιπόν το εξή. Μέχρι ε, πού, μέχρι σε ποιο βαθμό το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο θα είναι εργαλείο που θα εμβαθύνει τη δημοκρατική λειτουργία της Ένωσης και θα κάνει την Ευρωπαϊκή Ένωση να πλησιάσει τον Ευρωπαίο πολίτη. Μέχρι πού μπορούμε να φτάσουμε ε, με αυτό το στόχο. Αυτό είναι ένα πρώτο σχόλιο που θα ήθελα να κάνω. Διότι κύριε Ντομπρόφσκης, κύριε Επιτροπέ, ξέρετε, ε, ε, αναφερθήκατε σε τρεις παράγοντες επιτυχίας για το ευρωπαϊκό εξάμεινο και μιλήσατε για την ανακοίνωση και την επικοινωνία με τα εθνικά κοινοβούλια. Εγώ νομίζω ότι η επικοινωνία είναι πολύ μικρή, είναι αδύναμη με τα εθνικά κοινοβούλια. Τα εθνικά κοινοβούλια χρειάζεται να διαδραματίσουν πολύ πιο σημαντικό ρόλο κατά την ε, διενέργεια του ευρωπαϊκού εξαμήνου. Η κυρία Μαριάν Τάισεν μας υπενθύμησε ότι το εγχείρημα αυτό του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και το επαναλαμβάνω γιατί πρόκειται για εγχείρημα συντονισμού των οικονομικών και κοινωνικών πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, προχωράει. Εμείς όμως διαπιστώνουμε ότι υπάρχει ο Ευρωπαϊκός Πυλώνας για τα εργασιακά δικαιώματα, υπάρχει το βαθμολόγιο, σημαντικά όλα αυτά δεν λέω, όμως δεν έχουν τη θέση που τους αναλογεί. Ε, το Ευρωπαϊκό Κατόφλι ε, Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Εργασιακών Δικαιωμάτων θα πρέπει να ενισχυθεί στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Δεν είναι τόσο ηχηρό, δεν είναι τόσο εμφανές όσο θα έπρεπε. Είμαστε παραμονές του Brexit. Θα είναι σκληρό το Brexit, θα είναι ήπιο ή δεν θα υπάρχει συμφωνία για Brexit καθόλου. Όποια λύση και αν βρεθεί, σε κάθε περίπτωση το Brexit θα έχει αναγκαστικά αντίκτυπο στην καθημερινότητα, στη ζωή των πολιτών. Σε ποιο βαθμό λοιπόν ο αντίκτυπος του Brexit λαμβάνεται υπόψη στις πολιτικές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις πολιτικές προτεραιότητες του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Αυτά ήθελα να θέσω υπόψη. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο Πρόεδρος και εμείς σας ευχαριστούμε. Η κυρία Χίγκιν, Ιρλανδία, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Μίλησαν άλλοι γιατί, και άλλοι για την ανάγκη ενίσχυσης της φωνής των κοινοβουλίων και των εκπροσώπων τους ε, στην Ιρλανδία υπήρξε και μια εθνική συζήτηση για το θέμα αυτό. Πιστεύω όμως ότι θα πρέπει στον εθνικό διάλογο για τη διαδικασία του εξαμήνου να συμμετάσχει και η κοινωνία των πολιτών. Εμείς είχαμε στην Ιρλανδία νομίζω και είμαστε η μόνη χώρα μια τέτοια διάσταση του διαλόγου για το εξάμεινο Πιστεύουμε ότι αυτό είναι απαραίτητο έτσι ώστε να αναζωπηρωθεί και η συζήτηση με την κοινωνία των πολιτών για το τι κοινωνικό μοντέλο θέλουμε να έχουμε στο μέλλον και πώς μπορεί να ενταχθεί σε αυτό το κοινωνικό μοντέλο το ε, ε, εξάμεινο. Ε, επίσης, ε, πολύ συχνά ε, βλέπουμε ότι για την ανάπτυξη πολύ συχνά βάζουμε στόχους οι οποίοι είναι πάρα πολύ δύσκολοι και όταν μιλάμε ε, για θέματα όπως είναι ας πούμε οι σωστοί στόχοι, οι στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης, ε, αυτοί οι στόχοι θα πρέπει να επιτεχθούν ε, και σε σχέση και με το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο και λαμβάνοντας ε, υπόψη και το Brexit ε, ε, θα πρέπει να τα σκεφτούμε όλα αυτά και να τα δούμε μακροπρόθεσμα γιατί η ένταση και η πίεση μας κάνουν να σκεφτόμαστε λίγο βράχη πρόθεσμα και αυτό δεν είναι τόσο σωστό. Πιστεύουμε λοιπόν ότι θα πρέπει να ενισχυθεί ο διάλογος αλλά να ενισχυθεί και το κοινωνικό ο κοινωνικός ε, πυλώνας. Δεν είναι δυνατόν να λέμε ε, σε κάποιους δείκτες αν είναι κάτω από το μέσο όρο, πάνω από το μέσο όρο. Όχι, θέλουμε πραγματικά ποιοτικούς δείκτες και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σε εθνικό επίπεδο θα πρέπει οπωσδήποτε να έχουμε την δυνατότητα ε, να ε, ε, προσέχουμε και να στρέφουμε την προσοχή μας πάνω σε θέματα πριν γίνουν αυτά προβλήματα. Σας ευχαριστώ πολύ. Πιμένοφ από τους Σοσιαλιστικούς και Δημοκράτες της Λετωνίας. Θα μιλήσω αγγλικά. Η πιο μοδάτη λέξη είναι οι επενδύσεις. Και η μακροοικονομική σταθερότητα ήταν η πιο μοδάτη λέξη πριν από κάποια χρόνια. Φέτος είναι οι επενδύσεις για το ευρωπαϊκό εξάμεινο. Όσοι υπόσχονταν ότι τα, θα έρχονταν τα διεθνή κεφάλαια μόλις ε, υπάρξει οικονομική σταθερότητα διαψεύθηκαν επιβλήθηκαν πολιτικές δυσλιτότητες που οδήγησαν σε μεγάλη οδύνη στις κοινωνίες μας και φέρανε βιώσιμη τελμάτωση αντί για βιώσιμη ανάπτυξη στην οικονομία μας. Και τελικά δεν ήρθαν ποτέ οι επενδύσεις και τα, διεθνή, τα διεθνή κονδύλια. Οι εθνικές οικονομίες χρειάζονται δημόσιες επενδύσεις για να αυξηθεί η εσωτερική ζήτηση. Και για να έρθουν οι ιδιωτικές επενδύσεις θα πρέπει να προϋπάρχουν δημόσιες επενδύσεις, γιατί ο ιδιωτικός τομέας ακολουθεί τη ζήτηση. Η στρατηγική αναθεώρηση του Δημοσιονομικού Συμφώνου είναι απαραίτητη. Η μεθοδολογία για το προσδιορισμό του διαρθρωτικού αλήματος να επανεξεταστεί. Είναι μια πανεπιστημιακή μεταβλητή που είναι δύσκολο να υπολογιστεί και μπορεί να, δημιουργήσει, να οδηγήσει σε λάθη που στοιχίζουν πάρα πολύ στα κράτη-μέλη. Μία λύση θα ήταν να αντικατασταθούν οι διαρθρωτικές ισορροπίες με μία τιμή αξία δαπανών. Σε αντίθεση με τις διαρθρωτικές ανισορροπίες, η δαπάνη μπορεί να αντιμετωπιστεί πιο εύκολα. Από εκεί και πέρα, ο υπολογισμός της ενδυνάμει ανάπτυξης και του διαρθρωτικού ελλείμματος θα πρέπει να βασίζεται σε μεγαλύτερο ευρώ χρόνου και όχι μόνο στο διετέ ε, χρονικό περιθώριο που χρησιμοποιείται τώρα και η ευελιξία του Συμφώνου Σταθερότητας θα πρέπει να επεκταθεί απαλλάσσοντας την εθνική συγχρηματοδότηση των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών ταμείων και επενδυτικών ταμείων. Να απαλλαχθεί λοιπόν αυτό από ε, τον υπολογισμό για το έλλειμμα ε, και τη, δημοσιονομική ισορροπία. Ο κύριος Μπόργκη από το ΕΝΕΦ e και την Ιταλία. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ αγαπητέ συνάδελφοι και αγαπητοί συνάδελφοι. Uh, in the introductory remark... Uh, Στις εισαγωγικές παρατηρήσεις άκουσα διάφορες λέξεις όπως αξιοπιστία, οικειοποίηση, ιδιοκτησία, τέλεια. Αλλά αυτή η αξιοπιστία και αυτή η οικειοποίηση θα πρέπει οπωσδήποτε να μεταφραστούν σε ε, γεγονότα και σε στοιχεία. Στις εισαγωγικές ε, ε, παρατηρήσεις ε, η Ιταλία θεωρείται όσο μη συμμορφούμενη και έχω και μία εξαίρετη εδώ σελίδα όπου η Ιταλία ε, συμπεριλαμβάνεται στις χώρες οι οποίες έχουν υπερβολικό έλλειμμα. Αυτά είναι τα έγγραφα που μας δώσατε. Και με το βαθμολόγιο του 19. Και όλα αυτά δείχνουν ότι όμως ε, ε, τα πράγματα δεν είναι ακριβώς έτσι. Γιατί από τις 15 παραμέτρους η Ιταλία βρίσκεται πραγματικά κάτω από το μέσο όρο ε, της ε, παράβασης ας πούμε ή παραβίασης αυτών των στοιχείων υπάρχουν άλλοι που έχουν ε, τρεις παραβιάσεις, 7, 5, 3 κτλ. Η Ιταλία όμως μονάχα σε δύο παραμέτρους δεν είναι ε, καλός μαθητής ε, και ε, οι δύο αυτές παράμετροι είναι η ανεργία και το, το χρέος και οφείλεται η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι υποχρεώσεις που έχει επιβάλει Αυτά ευθύνονται, λέω, για το ότι οι παράμετροι αυτοί δεν γίνονται σεβαστές. Ε, αποτέλεσμα των ε, πολιτικών που έχουν επιβληθεί στην Ιταλία είναι η αύξηση του χρέους και της ανεργίας. Εγώ θα ήθελα να δω και άλλες παραμέτρους ε, σε, αυτόν το, σε αυτό το βαθμολόγιο αναφοράς. Ας πούμε, η χώρα που πληρώνει και η χώρα που δέχεται χρήματα από τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί είναι λίγο αστείο, είναι λίγο περίεργο να είναι σε μια χώρα που συμμορφούνται με τις περισσότερες παραμέτρους, μια χώρα που έχει πληρώσει από την αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωση και εξακολουθεί να πληρώνει, να τη δείχνουν με, τον, με το δάχτυλο από εκπροσώπους χωρών που μόνο υποδέχονται, συγγνώμη, υποδέχονται, μόνο δέχονται χρήματα. Αυτό σημαίνει ότι εδώ κάτι τρέχει. Και αν θέλουμε να είμαστε αξιόπιστοι πραγματικά, θα πρέπει με τον ίδιο τρόπο ακριβώς να φερόμαστε σε όλες τις χώρες, πράγμα που δεν συμβαίνει. Εάν δεν αρέσει σε κάποιους η χώρα ή η κυβέρνηση, τότε αρχίζει τα προβλήματα. Εάν αρέσει όμως η κυβέρνηση ή η χώρα, τότε αυτή η χώρα και αυτή η κυβέρνηση μπορούν να κάνουν τα πάντα. Ε, η χώρα, ας πούμε, του Επιτρόπου Μοσκοβισή περνάνε το 3% του ελλείμματος ε, ε, σε σχέση με το ΑΕΠ και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Ενώ η Ιταλία με 2% έλλειμμα σε σχέση με το ΑΕΠ ε, τη δείχνουμε με το δάχτυλο. Κάτι πρέπει να αλλάξει, γιατί διαφορετικά μη μου τσαμπουνάτε τώρα για την αξιοπιστία. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. συμφωνώ ε, αυτό που είπατε για τα στοιχεία και το βαθμολόγιο, για τα υπόλοιπα. Ε, εντάξει, καλό είναι που τα είπατε για να ζωντανέψει η συζήτηση για λίγο. Ε, στη συνέχεια θα αναφερθώ λίγο σε αυτό. Ο κύριος Βότσης από την Κύπρο, Σοσιαλιστές και Δημοκράτες. Αγαπητοί συνάδελφοι, η διαπίστωση ότι διαχρονικά έχουν επιτευχθεί ουσιαστικέ βελτιώσει στο ευρωπαϊκό εξάμεινο που συνέβαλαν στην απλοποίηση και την αύξηση τη αποτελεσματικότητά του είναι σωστή. Ταυτόχρονα είναι σωστή η επισήμαση ότι υπάρχει περιθώριο για περαιτέρω εξορθολογισμό και βελτίωση τη διαδικασία του ευρωπαϊκού εξαμήνου. Επί του παρόντο, τα χρονικά περιθώρια είναι ασφιχτικά και δρούν ανασταλτικά, αποθαρρύνοντα τη διεξαγωγή επικοδομητικού διαλόγου με την ενεργό εμπλοκή όλων των ενδιαφερομένων μερών σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Δράττουμε τη ευκαιρία να εκφράσω τι ανησυχίε μα ω προ τι πρόσφατε προσπάθειε που καταβάλλονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για ένταξη στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και συγκεκριμένα για συμπερίληψη στις ειδικέ αναχώρα συστάσει ζητημάτων που άπτονται του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού. Τέτοιε ενέργειες υποθάλπτουν τη διχόνοια και είναι αντίθετες προς τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που είναι η πρόθεση του κοινού καλού της Ένωσης και η καλλιέργεια πνεύματος αμοιβαίου σεβασμού, εμπιστοσύνης και ενότητας μεταξύ των Ευρωπαίων εταίρων. Η Κύπρος τάσσεται υπέρ της βελτίωσης της διαφάνειας και της λογοδοσίας για τα ζητήματα του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού, αλλά αποδοκιμάζει την επιχειρούμενη μετατόπιση τη αρμοδιότητα των ζητημάτων επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εκτιμούμε ότι το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο πρέπει να μείνει αυστηρά προσιλωμένο στου όρου εντολή του, ήτι το συντονισμό των οικονομικών, δημοσιονομικών και διαρθρωτικών πολιτικών των κρατών μελών τη Ένωση. Καταλήγοντα, θα ήθελα να τονίσω το ρόλο κλειδί που μπορούν να διαδραματίσουν τα εθνικά κοινοβούλια μέσω τη άσκηση επαρκού κοινοβουλευτικού ελέγχου τόσο κατά την διαμόρφωση των εθνικών μεταρρυθμιστικών προγραμμάτων και προγραμμάτων σύγκληση, όσο και κατά την παρακολούθηση τη υλοποίηση των ειδικών αναχώραση τάσεων, προκειμένου η διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου να επενδυθεί με εθνική κυριότητα και δημοκρατική νομιμοποίηση. Σα ευχαριστώ. Thank you. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Μάρδας, παρακαλώ, από την Ελλάδα και την Ευχαριστώ, Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε. Χρησιμοποιώντας τους εύστοχους όρους της κυρίας Τάισεν, ήθελα να σημειώσω αρχικά ότι εμείς ως Έλληνες δεν ανήκουμε στους βετεράνους των εξαμήνων, αλλά μάλλον στους νέους. Οπότε ε, θα ήθελα να θέσω μία ερώτηση η οποία μπορεί να φανεί πεζή και έχει ένα διαδικαστικό χαρακτήρα. Υπάρχει μία έκθεση ή ένας πίνακας έστω όπου στο πλαίσιο μιας επισκόπησης να φαίνονται οι παρεμβάσεις των κοινοβουλευτικών και από εκεί και πέρα ποια είναι η αντίδραση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με την έννοια που οδήγησαν αυτές οι παρεμβάσεις. Οδήγησαν στην ανάληψη κάποιας πρωτοβουλίας έτσι ώστε να εκπονηθεί κάποια μελέτη. Συνέβαλαν έτσι ώστε να έχουμε μία γνώμη, μία απόφαση, να έχουμε μία οδηγία ή έστω έναν κανονισμό. Ε, τι γίνεται σε ό,τι αφορά λοιπόν ε, όλο αυτό το διάλογο τον οποίο ζούμε όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Αν ε, ε, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο, έχω την αίσθηση ότι θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συντάσει ένα τέτοιο κείμενο ή έναν πίνακα, ο οποίος να διανέμεται ακολούθως στους συμμετέχοντες. Αν υπάρχει βέβαια, καθώς δεν τον έχουμε, καλό θα ήταν σε κάθε συνάντησή μας να, το, να τον είχαμε έγκαιρα. Ευχαριστώ πολύ. Thank you. Now, uh, Σας ευχαριστώ. Σίλβα Περέιρα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Σοσιαλιστές και Δημοκράτες. Uh, ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να συμφωνήσω κι εγώ με όλους ε, όσοι προηγουμένως αναφέρθηκαν στη σημασία του εξαμήνου και θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι η εργασία μας γίνεται στα πλαίσια μιας πρότασης της Κομισιόν που είναι πρόταση ανατολισμού των οικονομικών και δημοσιονομικών πολιτικών αυτό που ονομάζουμε ε, ετήσια επισκόπηση ανάπτυξης. Ευχαριστούμε την Κομισιόν για αυτήν την ισορροπημένη κατά την άποψή μου πρόταση που βασίζεται στους τρεις πυλώνες, που βασίζεται επίσης στις επενδύσεις, που υπεραμείνεται μεταρρυθμίσεων ε, οικονομικών ε, και συμπερίληψης, αλλά βεβαίως ε, αφορά και τα, την εξυγίανση το, την δημοσιονομική. Έχουμε ξεκινήσει να μελετούμε σε επικοδομητικό πνεύμα και πνεύμα συνεργασίας παρά ε, τις πολιτικές μας διαφορές. Ε, έχουμε αρχίσει λέω να μελετούμε το θέμα. Όμως ε, αναφέρομαι σε την επιβράδυνση η οποία φαίνεται να είναι πιο σημαντική από ό,τι θεωρούσαμε εκ πρώτης όψεως. Αυτό ισχύει για την Ιταλία. Η Γερμανία επίσης ε, από ό,τι φαίνεται μένει στάσιμη. Άρα ποιες είναι οι απαντήσεις που η δημοσιονομική και οικονομική πολιτική μπορεί να φέρει ε, σε αυτήν την κατάσταση. Ε, ε, θα πρέπει να γίνει κάποια τροποποίηση ριζική της οικονομικής, δημοσιονομικής πολιτικής και οπωσδήποτε θα πρέπει να διορθωθεί το έλλειμμα των επενδύσεων. Αυτό είναι μια έκκληση που πρέπει να απευθυνθεί σε όλες τις χώρες που έχουν την δυνατότητα να καλύψουν το έλλειμμα αυτό. Αυτό είναι πραγματικά σημαντικό εάν θέλουμε ε, να θεωρήσουν οι πολίτες ότι ε, η δημοσιονομική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης δίνει πραγματικές λύσεις. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Κρέτσου, ε, Σοσιαλιστές και Δημοκράτες από τη Ρουμανία. Thank you very much. Dear colleagues... Ευχαριστώ πολύ. Αγαπητοί συνάδελφοι, έχουμε τρία βασικά εργαλεία παρέμβαση σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να πετύχουμε του στόχου μα. Το ένα είναι το νομοθετήν, δηλαδή να έχουμε κοινή νομοθεσία. Το δεύτερο είναι το να χρηματοδοτούμε μέσα από τον προπολογισμό και συνδεδεμένα χρηματοπιστωτικά εργαλεία. Και το τρίτο είναι ο συντονισμό, να συντονίζουμε τι εθνικέ πολιτικέ κατά τη διάρκεια του ευρωπαϊκού εξαμήνου. Το πιο ασθενέ, το πιο αδύναμο εργαλείο είναι ο πολιτικός συντονισμό. Θα μπορούσε να είχε λειτουργήσει αν είχαμε ως αντιστάθμισμα ισχυρή πολιτική βούληση για να το πράξουμε. Δεύτερον, την ίδια πολιτική βούληση παντού, δηλαδή ίδιοι στόχοι, ίδια δυνατότητα, ίδια διοικητική ε, διοικητικό δυναμικό και προπολισμό για την υλοποίηση των πολιτικών και τρίτον ε, συστάσεις που να έχουν συνέπεια και συνοχή μεταξύ τους. Αν τα είχαμε αυτά θα το είχαμε καταφέρει και θα το είχαμε ενισχύσει ως εργαλείο. Τώρα έχουμε μια άτυπη έγκριση χωρίς ε, σαφείς συνέπειες σε ό,τι αφορά την υλοποίηση. Η πολιτική βούληση είναι ασθενής. Οι κυβερνήσεις εκπροσωπούν διαφορετικές κατηγορίες πολιτικών συμφερόντων και έχουν να αντιμετωπίσουν ιδιαίτερη πραγματικότητα, ιδιαίτερες συνθήκες σε, κάθε, σε κάθε κράτος μέλος. Τα κράτη-μέλη κάνουν τις δικές τους διαγνώσεις για, τη, για το δικό τους κοινωνικό ιστό και θέτουν προτεραιότητες σε εθνικό επίπεδο. Ε, ναι, μερικές φορές η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει και το Συμβούλιο εγκρίνει ειδικέ συστάσεις αναχώρα για το ίδιο το κράτος μέλος, το οποίο αντί να συγκλίνει ουσιαστικά κινήθηκε προς την αντίθετη κατεύθυνση και υπονόμευσε τη θέση του άλλου κράτους μέλους και αντιστρόφως. Και όταν ρώτησα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή γιατί υπάρχει αυτή η ασυνέπεια, ε, είχα διαφορετικές απαντήσεις γιατί είχαμε ανθρώπους από διαφορετικές γενιές να προείστανται των διαφορετικών γενικών διευθύνσεων και γι' αυτό ήταν τόσο ποικίλε οι απαντήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έχουμε συστάσεις για λιτότητα από τη Γενική Διεύθυνση για τα Οικονομικά και συστάσεις για, το για την καταπολέμηση της φτώχειας και των ανισοτήτων από τις Γενικές Διευθύνσεις που υπάγονται στην Επίτροπο κυρία Τάισεν. Άρα, οι συστάσεις για το οικονομικό σκέλος έχουν εφαρμοστεί κατά 85% και οι συστάσεις για την εκπαίδευση και τις κοινωνικές πολιτικές έχουν τεθεί στο περιθώριο. Μόνο 7% είναι το ποσοστό υλοποίησης. Για το 2018, εκτός από τις συστάσεις που περικόπτουν τα υφιστάμενα δικαιώματα. Πρέπει να γνωρίζουμε λοιπόν αυτές τις δυσκολίες του συντονισμού και να αναλάβουμε δράση. Ιδαλλιώς, πολύ λένε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη κάνει το καθήκον της και γι' αυτό έχει έρθει η ώρα να αποχωρήσει από το προσκήνιο. Θα ήταν κρίμα αυτό μεγάλο και θα ήταν και κίνδυνος μεγάλος, γιατί σημαίνει ότι θα έχουμε ξεχάσει πόσο σημαντική είναι η ειρήνη και η συνεργασία για να πετύχουμε το σημερινό επίπεδο ανάπτυξης. Χάρη στην ειρήνη που έφερε η Ευρωπαϊκή Ένωση πετύχαμε αυτό το επίπεδο ανάπτυξης και δεν πρέπει να το ξεχνούμε αυτό. Χαίρομαι όμω, διότι με, την, με το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο έχουμε ξεκινήσει έναν ισχυρό διάλογο μεταξύ Ευρωπαϊκών Θεσμικών Οργάνων και Κρατών Μελών και μεταξύ ημών όλων. Αυτό είναι μια καλή βάση για να χτίσουμε πολιτικές καλύτερε με περισσότερη συνέπεια και συνοχή μεταξύ τους που θα ωφελήσουν ακόμη περισσότερο του πολίτε στο μέλλον. Ευχαριστώ. Όλγα Ζερίχεν, πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων από Πλευρά Επιτροπή των Περιφερειών. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι αγαπητοί συνάδελφοι. Καταρχάς, ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για την πρόσκληση. Για άλλη μια φορά μας καλέσατε στη διάσκεψη αυτή για να εκπροσωπήσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών. Οι εκθέσεις αναχώρα που θα δημοσιεύσει την άλλη εβδομάδα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μα δώσουν μια εικόνα για το πώς έχουν εφαρμόσει τις στάσεις οι διάφορε χώρες τους τελευταίους μήνες. Υπάρχει γενική αίσθηση ότι μετά την κρίση οι διαρθωτικές μεταρρυθμίσεις ε, ε, προχωρούν ε, με βραδείς ρυθμούς, γιατί ακριβώς δεν το έχουν κάνει κτήμα τους αυτό τα κράτη-μέλη. Νομίζουμε ότι δεν έχουν καταβληθεί αρκετές προσπάθειες για να κατανοήσουμε γιατί δεν έχει γίνει κτήμα των κρατών και γιατί δεν είναι αποτελεσματική η απάντηση. Είναι όμως σημαντικό να έχουμε την απάντηση αυτή, γιατί έχουμε δύο νέα στοιχεία ε, που αυξάνουν τη σημασία του οικονομικού εξαμένου. Πρώτο καινούριο, ένα πρόγραμμα υποστήριξης των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Φαίνεται να έχει πιστεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι το πρόβλημα είναι ε, η κατάσταση στην οποία βρίσκονται τα δημόσια οικονομικά. Ε, ε, πράγμα που δεν επιτρέπει τη στήριξη των ομάδων που πλήττονται από τις μεταρρυθμίσεις. Ήμουν εισηγήτρια στην Επιτροπή Περιφερειών, η οποία διαφωνεί όμως με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εμείς θεωρούμε ότι οι συστάσεις αναχώρα για τις μεταρρυθμίσεις δεν έχουν γίνει κτήμα των κρατών για το λόγο ότι αυτά καταρτίζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά από συνεννόηση ε, με τις εθνικές κυβερνήσεις, ε, χωρίς συμμετοχή στις περισσότερες περιπτώσεις των αρχών της τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης, με εξαιρέσει στις ομοσπονδιακές χώρες και χώρες που έχουν μακρά παράδοση συνεργασίας των διάφορων επιπέδων ε, διακυβέρνησης. Αλλά δεν ισχύει παντού αυτό. Θυμίζω, όπως είχε πει και τον Οκτώβριο του 2018 στην έκθεσή της για την επικουρικότητα Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η ΟΤΑ και οι περιφερειακές αρχές δεν συμμετέχουν. Αλλά εκείνες καλούνται όμως να υλοποιήσουν σε πολλές περιπτώσεις την ευρωπαϊκή νομοθεσία και γνωρίζουν περισσότερο από τον καθένα τις ανάγκες ε, της περιφέρειας και έρχονται σε άμεση επαφή με τους πολίτες. Πρέπει λοιπόν να συμμετέχουν στο ευρωπαϊκό εξάμεινο ε, βάσει της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης και της εταιρικής σχέσης από την αρχική φάση, από τη στιγμή που εντοπίζονται οι μεταρρυθμίσεις που πρέπει να γίνουν. Αν συνέβαινε κάτι τέτοιο θα είχαν πολύ μεγαλύτερη ε, ευστοχία οι συστάσεις και θα μπορούσαν να εφαρμόζονται καλύτερα. Και το δεύτερο είναι πιο στενή σχέση τώρα με την πολιτική συνοχής. Μακροπρόθεσμες επενδύσεις χρειάζονται από τα κράτη-μέλη Ποιε θα είναι οι επενδύσεις αυτές. Οι συστάσεις του εξαμήνου 2019 αναφέρονται στη συνοχή για το διάστημα 2021-2027. Η πολιτική συνοχή ήδη βασίζεται στην πολυεπίπεδη διακυβέρνηση και στην εταιρική σχέση και θα πρέπει να παραμείνει. Περιορίζεται όμως από το ευρωπαϊκό εξάμεινο. Και αυτό θα ε, προκαλούσε ένα μεγάλο πρόβλημα ε, επικουρικότητας και δεν βοηθάει ε, να υιοθετήσουν και να ενστερνιστούν τις μεταρρυθμίσεις στα κράτη-μέλη. Ο Πρόεδρος διακόπτει την ομιλήτρια. Τον Απρίλιο η Επιτροπή των Περιφερειών θα εγκρίνει μια νέα γνωμοδότηση για τη σχέση πολιτικής συνοχής με το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο και θα ζητήσει από την Ευρωπαϊκή, την Προεδρία μάλλον του Συμβουλίου, τη Ρουμανική, να ετοιμαστούν οι πόλεις και οι περιφέρειες να αντιμετωπίσουν τις ανάγκες τους με τρόπο ευέλικτο. Ευχαριστώ και σας εύχομαι καλή συνέχεια των εργασιών σας. Uh, ε, Mr. Ευχαριστώ πολύ ο κύριος Βρομπλεύσκη, ECR ε, ε, από την Πολωνία. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Βεβαίως είναι σαφή τα πλεονεκτήματα ε, της, ε, του εξαμήνου αλλά υπάρχουν και λήψεις ε, τις οποίες διαπιστώνουμε σε σχέση με το μη ικανοποιητικό επίπεδο υλοποίησης των συστάσεων από τις διάφορες χώρες ενδεχομένως γιατί δεν υπάρχουν οι μηχανισμοί υποστήριξης έτσι ώστε να υλοποιηθούν οι μεταρρυθμίσεις που έχει ζητήσει από τις χώρες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, στα πλαίσια των ε, συζητήσεων ε, βέβαια για τον προϋπολογισμό θα πρέπει να συζητηθούν τα θέματα αυτά και στα πλαίσια και των συζητήσεων για το ΠΔΠ μέχρι το 2027 θα πρέπει σίγουρα να ληφθεί υπόψη η ανάγκη να μην πειράξουμε τους πόρους συνοχής. Είναι σημαντικό επίσης ε, και πριν ακόμα ε, δημοσιοποιηθούν οι συστάσεις ε, η Κομισιόν έρχεται σε επαφή με τις χώρες έτσι ώστε να είναι καλύτερη η επαφή με τις χώρες αλλά και καλύτερος και ο βαθμός υλοποίησης από τις χώρες μέλη. Εμείς είμαστε ανοιχτοί να συνειζητήσουμε το ενδεχόμενο κινητροδότησης των επενδύσεων, των ε, διαρθρωτικών επενδύσεων αλλά όλα αυτά δεν θα πρέπει καθόλου να αποδυναμώσουν την υφιστάμενη πολιτική συνοχής. Όλα αυτά βεβαίως είναι πάρα πολύ σημαντικά έτσι ώστε ε, η πρόοδος όσον αφορά ε, τα διαρθρωτικά να είναι ίδια σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Μπανιάη από την Ιταλία και το ΙΕΝΕΦ. E Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, πολλοί συνάδελφοι υπογράμμισαν ότι θα πρέπει να είναι σε μηχανισμό συντονισμού το εξάμεινο. Εγώ δεν το δέχομαι ακριβώς ε, και αναρωτιέμαι για ποιο σκοπό ε, συντονίζουμε τις ε, πολιτικές μας για να μειωθεί ας πούμε το δημοσιονομικό έλλειμμα, για να έχουμε ευημερία, για να έχουμε μεταρρυθμίσεις ή ανάπτυξη. Εάν ε, συγκρίνουμε την, την ε, ανάπτυξη της ε, Ευρωζώνης με άλλα, άλλα μεγάλα μπλοκ της παγκόσμιας οικονομίας, διαπιστώνουμε ότι δεν έχει δώσει και πολλά αυτός ο μηχανισμός και άλλωστε πρόκειται για ένα μηχανισμό ο οποίος δεν είναι διαφανής και λειτουργεί με τρόπο περίεργο και όχι πάντα ικανοποιητικό. Επίσης ε, δεν λαμβάνονται υπόψη όλα τα στοιχεία που θα έπρεπε να ληφθούν ε, έτσι ώστε το βαθμολόγιο να έχει πραγματική έννοια. Μονάχα ορισμένες οικονομικοί, οικονομικοί παράμετροι λαμβάνονται ε, υπόψη και ας πούμε ένας δείκτης όπως είναι το ισοζύγιο δεν λαμβάνεται υπόψη ο, ως μηχανισμός λοιπόν ε, συντονισμού μεταξύ των ευρωπαϊκών οικονομικών στρατηγικών ε, δεν είναι τόσο ικανοποιητικός και πιστεύω μάλιστα ότι μπορεί να αποτελέσει και με σαφή απειλή ε, ανάμεσα ας πούμε όσον αφορά την οικονομική πολιτική και τις σχέσεις ανάμεσα σε εμά, ας πούμε, και τις ε, Ηνωμένε Πολιτείε, ε, κυρίως λαμβάνοντας υπόψη και στοιχεία όπως είναι το εξωτερικό ε, χρέος. Παρατηρήσεις, λοιπόν. Στο εγγύς μέλλον πιστεύουμε ότι η Ευρώπη θα πρέπει να λάβει το θέμα του συντονισμού πολύ στα σοβαρά και για το σκοπό αυτό ένα από τα πιο σημαντικά, ε, σημαντικό είναι ότι οι φορολογικοί κανόνες ε, θα πρέπει να ε, ρυθμίζονται, να σχεδιάζονται καλύτερα. και να υπάρχει ακαιρεότητα όσον αφορά τους υπολογισμούς και όσον αφορά τις συστάσεις που γίνονται στις χώρες. Ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Τελευταίος ο μιλητής, Ιάνν Ντεμελένα, η συγγήτρια της γνωμοδότησης της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής. Τρία λεπτά, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς θέλω να σας ευχαριστήσω γιατί επιτρέψατε στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή να πάρει το λόγο μέσω εμού και να εκφραστεί ενώπιόν σας. Έχουμε συντάξει μια γνωμοδότηση για την ετήσια εξέταση της ανάπτυξης για το 2019 που θα ψηφιστεί στη Σύνοδο της Ολομέλειάς μας τις επόμενες μέρες. Τι περιέχει η γνωμοδότησή μας. Πρώτον, την εξή διαπίστωση. Ε, μπροστά στις αμφιβολίες και αβεβαιότητες και σε ευρωπαϊκό και σε παγκόσμιο επίπεδο και με βάση την οικονομική επιβράδυνση είναι απαραίτητο να ξαναξεκινήσει η οικονομία μέσω των επενδύσεων και μέσω της αύξησης της παραγωγικότητας. Είναι ανάγκη να μειωθούν οι κοινωνικές ανισότητες με το ευρωπαϊκό ελάχιστο κατόφλι εργασιακών δικαιωμάτων που θα πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του ευρωπαϊκού εξαμήνου. Μία προσθήκη που δεν θα πρέπει να παραμελεί κανείς είναι το γεγονός ότι θα άρμοζε και θα τέριαζε να αντιμετωπίσουμε την κλιματική αλλαγή μειώνοντας την εξάρτηση της οικονομίας από τον άνθρακα. Αυτή η ετήσια εξέταση του ρυθμού ανάπτυξης είναι μια πολύ μεγάλη και σημαντική άσκηση βιώσιμης ανάπτυξης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και γι' αυτό θέλουμε να ε, το βαφτίσουμε το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο ετήσια εξέταση της βιώσιμης ανάπτυξης. Θέλουμε να του αλλάξουμε την ονομασία δηλαδή. Σε αυτή τη διαδικασία οι κοινωνικοί εταίροι η οργανωμένη κοινωνία των πολιτών είναι ένας πολύ σημαντικός εταίρο. είναι συνεργάτες πάρα πολύ σημαντικοί και πρέπει να του λαμβάνουμε υπόψη και να μην ξεχνούμε την πραγματικότητα επιτόπου. Μια άλλη παρατήρηση έχει να κάνει με τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Είναι πολύ σημαντικό οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις να εντοπίζονται καλύτερα, να διευκρινίζονται περισσότερο, διότι μεταξύ των στόχων έναρξη και των ε, επιτευγμάτων επιτόπου η απόσταση είναι μεγάλη και η απόκληση, η συχνά είναι μεγάλη. Είναι συχνό η συχνή ανάγκη να μπορούμε να τους αξιολογήσουμε στη συνέχεια, τις μεταρρυθμίσεις να τις αξιολογούμε για να μην διαπράττουμε λάθη. Προσοχή να δώσουμε στον επίγοντα χαρακτήρα ορισμένων κοινωνικών δράσεων. Έχουμε κοινωνικές ανισότητες που όλο και οξύνονται εντός των κρατών μελών ή μεταξύ των κρατών μελών. Και την απάντηση θα βρούμε από τη μία στη μισθολογική στήριξη. Σε πολλές χώρες η εξέλιξη των μισθών είναι λιγότερη από την εξέλιξη της παραγωγικότητας και αυτό έχει αντίκτυπο αρνητικό στο κόστος ζωής. Το μισθολόγιο, η μισθή είναι ένα εργαλείο στήριξης της εσωτερικής αγοράς και ένα εργαλείο αναθέρμανσης τη οικονομίας. Μιλήσαμε για το ποσοστό απασχόλησης που βαίνει αυξανόμενο. Να μην ξεχνάμε όμως ποια είναι η ποιότητα αυτών των νέων θέσεων απασχόλησης που δημιουργούνται. Το 2007, το 2017 ο αριθμός των ωρών που δούλεψε κανεί και που προσφέρει τη δούλεψή του για αυτές τις ώρες είναι μικρότερο από τον αντίστοιχο του 2016. Άρα έχουμε όλο και πιο αβέβαιες θέσεις απασχόλησης και αυτό είναι πρώτο πρόβλημα. Πρέπει να έχουμε δίκαιη φορολογία με βάση τη φοροδοτική ικανότητα του πολίτη. Έγινε λόγο και για τα δημόσια οικονομικά. Είναι πολύ καλό να τα πετυχαίνουμε όλα αυτά με αντικυκλικές μακροοικονομικές πολιτικέ, όμω έχουμε και το χρυσό κανόνα που ε, ε, αποκλείει από το σύμφωνο σταθερότητας τη δημόσιες επενδύσεις υψηλής προστιθέμενη αξία. Όλα αυτά λοιπόν αξίζει να τα σκεφτούμε και να τα λάμε πολύ σοβαρά υπόψη. Ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ να δώσω το λόγο στα μέλη του Προεδρείου του πάνελ για σχόλια και απαντήσεις. Κύριε Ντομπρόφσκης, Αντιπρόεδρε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Γκουαλτιέρη, αξιότιμοι συνάδελφοι. Πολλές ερωτήσεις ε, έγιναν, όπως και σχόλια. Θα προσπαθήσω να επανέλθω και να απαντήσω ε, ομαδοποιώντας ε, λίγο τις ερωτήσεις ανάλογα με το θέμα. Καταρχάς, το θέμα της εφαρμογής των συστάσεων αναχώρα και των επιδόσεων σε αιτήσια βάση των κρατών μελών αν ε, πραγματικά εξετάσουμε ε, ετησίως ε, την εφαρμογή, δεν είναι τόσο ικανοποιητική, γιατί οι μεταρρυθμίσεις χρειάζονται χρόνο. Αν το δούμε σε βάθος χρόνου, καταλαβαίνουμε ότι εφαρμόζονται πολύ καλύτερα. Τώρα λοιπόν επεξεργαζόμαστε το εξάμεινο για να δούμε πώς μπορεί να βελτιωθεί αυτή η εφαρμογή και διαφαίνονται δύο νέα στοιχεία και έννοιες, το είπαν και πολλοί συνάδελφοι. Ε, πώς συνδέεται η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση με το ευρωπαϊκό εξάμεινο. Ήδη από το τρέχον εξάμεινο και τις φετινές εκθέσεις αναχώρα ε, ε, έχουμε ένα παράρτημα που έχει να κάνει με τις επενδύσεις, τα σχέδια και τις προτεραιότητες των επενδύσεων που συνδέονται με το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Θέλω να τονίσω ότι δεν ε, μπορούμε να έχουμε μία ενιαία λύση με ε, αντιγραφή ε, κάποιων σχημάτων και μεταφορά τους άλλου. Οι επενδύσεις χρειάζονται και χρειάζεται και υποστήριξη για να επιτευχθεί η σύγκληση. Ε, υπάρχει ο κανονισμός των κοινωνικών ε, διατάξεων και κάποια άλλα νομοθετήματα ε, τα οποία θα μας απασχολήσουν ως προς την αναλογικότητα, την προσθετικότητα και τη συμπληρωματικότητα. Έγινε μεγάλη αναφορά επίσης και στην κοινωνική διάσταση του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Τα τελευταία δύο χρόνια περίπου έχουμε ενισχύσει την κοινωνική διάσταση και συμπεριλαμβάνουμε το κοινωνικό βαθμολόγιο, αλλά ε, ε, παρακολουθούμε και την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων διά του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Ε, Στι συστάσει αναχώρα, το 1 τρίτο περίπου των συστάσεων έχει να κάνει με τι προτεραιότητε παιδεία και κοινωνικών θεμάτων. Θα εξακολουθήσουμε να εργαζόμαστε προ την κατεύθυνση αυτή γιατί όπως λένε και τα έγγραφα για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο, συμπεριλαμβανομένης και της πολιτικής και των ε, βασικών μας προτεραιοτήτων, τι λέμε, ότι δεν αρκεί να έχουμε οικονομική μεγέθυνση, αλλά ανάπτυξη της οικονομίας χωρίς αποκλεισμούς. Ε, δηλαδή θα πρέπει να αντιμετωπίζουμε τις ανισότητες ε, αναδιανομής ε, του εισοδήματος. Έγινε λόγος επίσης για τους δημοσιονομικούς κανόνες και πώς αυτοί συνδέονται με τις επενδύσεις. Το συζητούμε αυτό παγίως. Ήδη από το 2015 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εκδώσει ανακοίνωση για τη βέλτιστη χρήση ε, της ευελιξίας στο Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης, όπου αναφέρουμε αυτό το στοιχείο των επενδύσεων. Ε, προσωρινά επιτρέπουμε στα κράτη-μέλη να αποκλίνουν από τους δημοσιονομικούς στόχους εάν υπάρχουν επενδύσεις ε, και συγχρηματοδότηση ε, από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και υπάρχουν χώρες που επωφελήθηκαν από τη συγκεκριμένη ρήτρα. Ε, σε ό,τι αφορά τώρα τον ισοσχεδιασμό του προϋπολογισμού, έσοδα, δαπάνες, Όλα αυτά είναι θέματα που έχουν να κάνουν με το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο και που λαμβάνει υπόψη το, το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Έχουμε συστήσει σε κάποιες χώρες ε, να χρησιμοποιήσουν ε, τα πλεονάσματα που έχουν ε, για να τονώσουν τις επενδύσεις και τη ζήτηση. Παράδειγμα, η Γερμανία και κάτω χώρες. Οι δύο αυτές χώρες επίσης αντιμετωπίζουν μικρονομικές ανισορροπίες γιατί έχουν πάρα πολλά πλεονάσματα ε, πάνω από 6% ε, ε, του ΑΕΠ. Πλεόνασμα τραξιών συναλλαγών. Όλα αυτά λαμβάνονται υπόψη στο Ευρωπαϊκό Εξάμεινο και στη σύσταση. έγιναν κάποιες ερωτήσεις ειδικά σχετικά με τις δημοσιονομικές ε, επιδόσεις στην Ιταλία. Ακούστηκε το 2% έλλειμμα. Μα ακριβώς αυτό ε, το έλλειμμα μειώθηκε στο 2% μετά τις συζητήσεις που είχαμε εμείς με τις Ιταλικές αρχές. Και γι' αυτό δεν ανοίξαμε τη διαδικασία υπερβολικού λύματος και σε σχέση με το χρέος. Στην περίπτωση της Ιταλίας υπάρχουν μακροοικονομικές ανισορροπίες λόγω του υψηλού δημοσίου χρέους. Είναι το δεύτερο χρέος ε, προς το ΑΕΠ ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση από όλα τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αφορά και τον τραπεζικό τομέα αυτό. Η Ιταλία έχει από τα υψηλότερα επίπεδα μη εξυπηρετουμένων κόκκινων δανείων ε, από όλα τα κράτη-μέλη. αν δεν απατώμε, είναι πολύ ψηλό. Ε, και αυτές οι ανισορροπίες και του προπολογισμού θα πρέπει να ε, αντιμετωπιστούν για να μην αυξάνεται το έλλειμμα αντί να μειώνεται γιατί αυτό μπορεί να οδηγήσει σε αστάθεια, σε αύξηση των επιτοκίων, σε μείωση των δικτών εμπιστοσύνης πράγμα που θα έχει αρνητικές επιπτώσεις γενικότερα και στις επενδύσεις. Ως αποτέλεσμα όλων αυτών δεν είναι απορία άξιο που η επιβράδυνση στην Ιταλία ήταν πολύ πιο έντονη από ό,τι σε οποιαδήποτε άλλη χώρα. Και ε, σύμφωνα με την ε, χειμερινή πρόβλεψη, η Ιταλία σήμερα αναπτύσσεται με τους χαμηλότερους ρυθμούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά. Ε, θέλω να ευχαριστήσω όλους τους βουλευτές για τη συμμετοχή σας. Έγιναν πολλές προτάσεις για μεγαλύτερη συμμετοχή και ισχυρότερη και των Εθνικών Κοινοβουλίων στο Ευρωπαϊκό Εξάμεινο ε, ε, Ευρωπαϊκή Κοινοβουλευτική Εβδομάδα είναι μια καλή φόρμουλα να συμμετέχουν περισσότερο τα Εθνικά Κοινοβούλια και να έρχεται σε επαφή και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τα Εθνικά Κοινοβούλια, πράγμα που γίνεται έτσι κι σε τακτά χρονικά διαστήματα. Ευχαριστώ. Thank you. Thank you, Mr. Chairman. Well, President... Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ο Πρόεδρος Γκουελκέρη μου ζήτησε ε, να είμαι σύντομη και αυτό θα κάνω. Νομίζω ότι ε, μπορούμε να πούμε ότι πέρσι κυρίως προσπαθούσαμε να δούμε με ποιο τρόπο θα καταφέρουμε να ξεπεράσουμε ε, και τα τελευταία στοιχεία της ε, κρίσης. Γιατί είναι γεγονός βέβαια ότι ζούμε σε κόσμο που αλλάζει γρήγορα και διαρκώς και πολλοί στρέφονται προς εμάς, οι πολίτες στρέφονται προς εμάς για να δουν ποιες αλλαγές ε, θα κάνουμε αυτά, τα λαμβάνουμε υπόψη μας ε, στο εξάμεινο. Δεν ε, πρόκειται να κάνω μία ακόμα ανάλυση. Θα προσπαθήσω να απαντήσω τις ερωτήσεις, τις ερωτήσεις σας, αλλά το σημαντικό είναι τα, οι δεξιότητες, τα κοινωνικά θέματα, αυτά τα σημεία να τα τονίσουμε και να τα υποστηρίξουμε. Ε, βέβαια υπάρχουν και πολλές αρμοδιότητες οι οποίες βρίσκονται στα χέρια των περιφερειών, των τοπικών κοινωνιών ε, και ε, βέβαια εδώ δεν θα αναλύσουμε ποιος είναι υπεύθυνο γιατί, α, απλώς να πούμε ότι πολλά πρέπει να γίνουν και πρέπει να τα κάνουμε μαζί διαβλέπω ότι έχετε παρατηρήσεις ε, σχετικά με την ε, ένταξη του κοινωνικού πυλώνα. Σας είπα όμως ότι έχουμε πολλές, πολύ περισσότερες ε, συστάσεις αναχώρα κοινωνικού περιεχομένου από ότι τις ε, προηγούμενες ε, χρονιές. Ε, ναι, είναι γεγονός ότι η Κομισιόν θέλει όλος αυτός ο μηχανισμός, όλη αυτή η άσκηση να αποκτήσει μεγαλύτερο κοινωνικό πρόσημο σε σχέση με το βαθμολόγιο. Ναι, βασιζόμαστε και στο βαθμολόγιο αλλά και στους στόχους του 2020. Θα πρέπει τώρα να προβλέψουμε το τι θα κάνουμε μετά και να αναπτύξουμε ένα νέο πλαίσιο το οποίο θα ανταποκρίνεται ε, στους ε, ε, στόχους βιώσιμης ανάπτυξης και κοινωνικής ανάπτυξης του 2030. Αναφέρεται ότι τα τα ταμεία θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για τις μεταρρυθμίσεις για την ανάπτυξη των περιοχών, ναι, και το ΠΔΛΤΑΠ θα χρησιμοποιηθεί και για να καταρτιστούν λειτουργικά προγράμματα πιο εμπνευσμένα από ό,τι στο παρελθόν. Ορισμένα μεταξύ μόνο αναφέρατε το γεγονός ότι έχουμε ψηλότερα ποσοστά απασχόλησης, ε, συμφωνώ, αλλά δεν είναι πάντα όλες οι θέσεις και το σύνολο της απασχόλησης ποιοτικό. Ε, θα πρέπει να το δούμε αυτό. Θα ε, υπάρχουν επίσης ε, άτυπα, μη τυπικά συμβόλαια, συμβάσεις που εθελοντικά πολλές φορές βέβαια επιλέγουν και οι εργαζόμενοι και είναι πιο ευέλικτα. Εμείς αρχίζουμε να ε, εφαρμόζουμε όλες τις αρχές βάσει και των νομοθετικών προτάσεων και υπάρχει ας πούμε ε, το κείμενο για τις ε, διαφανείς και προβλέψιμες συνθήκες εργασίας που αφορά κυρίως και μπορεί να βοηθήσει ανθρώπους σε άτυπες ε, συμβατικές ε, μορφές. Επίσης έχουμε κάνει και μία πρόταση σύσταση στα κρατημέλη όσον αφορά την πρόσβαση για όλους στην, ε, στην κοινωνική ασφάλιση. Άκουσα και κάποιες παρατηρήσεις για τους μισθούς. Βεβαίως και αυτό εμείς στις παρατηρήσεις αναχώρα για ορισμένες χώρες έχουμε αναφέρει ότι υπάρχει δυνατότητα, υπάρχει περιθώριο Αύξηση βελτίωση των μισθών, αλλά καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν μπορεί να λυθεί στα πλαίσια του εξαμήνου. Είναι ένα θέμα των κοινωνικών εταίρων και των χωρών. Αυτά γιατί δεν θέλω να μακρηγορήσω, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι η συζήτηση ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και ελπίζω να τη συνεχίσετε και αύριο στον ίδιο τόνο. Νομίζω ότι όλοι εμείς συμφωνούμε πάνω στο γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Εξάμενο είναι ένα γεγονός εξαιρετικά σημαντικό, κρίσιμη σημασίας και ε, θα μπορούσε να αποδώσει πολύ περισσότερα, να αξιοποιήσει περισσότερο το δυναμικό του. Και αυτό δεν μας εκπλήσει γιατί το εγχείρημα συντονισμού εθνικών οικονομικών πολιτιών χωρίς ε, σαφή διαμοιρασμό των αρμοδιοτήτων με στη συνθήκη και με την ε, δημοσιονομική εποπτεία του προϋπολογισμού μόνο είναι ένα πολύ περίεργο εγχείρημα. Τα ομοσπονδιακά κράτη δεν έχουν να το κάνουν ε, έτσι. Έχουν πολύ πιο απλή διαδικασία γιατί υπάρχει ομοσπονδιακός προπολογισμό και η περιφερειακή των εκάστοτε πολιτιών. Από εκεί και πέρα. Αν θέλουμε να δούμε στην πράξη πώς έχει λειτουργήσει το ευρωπαϊκό εξάμεινο αυτά τα χρόνια, σίγουρα ε, βλέπουμε ότι ε, είχε βελτιωμένες επιδόσεις. Δεν λέω απαραίτητα ότι τα αποτελέσματα ήταν πιο καλά. Λέω ότι Έχουμε ένα ισχυρό επίπεδο δεσμευόμενου συντονισμού. Πολλοί πιστεύουν ότι αυτό λειτουργεί αμφίδρομα. Πιστεύω ότι το 2011, 2012, 2013 και 2014 η δημοσιονομική εποπτεία και ο συντονισμός των οικονομικών πολιτικών πέτυχαν. Όμως, εάν έχουμε ένα κακό μείγμα οικονομικής πολιτικής ή όχι το βέλτιστο δυνατό, αν έχουμε για παράδειγμα διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που ουσιαστικά δόθηκαν σε δύο εταιρείε και έχουμε εσωτερική υποτίμηση και cross-cutting, πρέπει να πω ότι ως Επιτροπή εμείς προσπαθήσαμε να υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία, να ε, έχουμε κοινωνική διάσταση, να έχουμε πιο ισορροπημένο μείγμα πολιτικής. Έχω προσπαθήσει αυτό στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και νομίζω ότι έχουμε δει πολύ καλύτερα αποτελέσματα και οφείλουμε αυτό να το αναγνωρίσουμε. Δεν είναι κάποιοι κακοί και κάποιοι άλλοι ή κακοί ή καλοί. Ξέρετε κύριε Μπόρκη, δεν είναι το ύψος του ελλείμματος σε ονομαστική αξία. Ε, το θέμα είναι ποιες αλλαγές θεσπίζει ο νέος προϋπολογισμός. Εάν έχετε ε, ένα σχέδιο, είναι άνευ η διαρθρωτική μείωση του 0,6% και χάρη στην ευελιξία ο λίγων εξημών έχουμε συμφωνία με την Ιταλία που θα έχουμε ε, ε, μείωση 0,2% διαρθρωτική μείωση. Άρα η ευελιξία δεν λαμβάνεται υπόψη στη διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος. Επομένως, θεωρώ ότι είναι θετική έκβαση, παρόλο που ασκήθηκε κριτική για το περιεχόμενο αυτού του προϋπολογισμού. Αλλά ας μην γίνει συζήτηση για τα ενδοϊταλικά θέματα. Δεν θα πω λοιπόν ότι μέχρι τώρα όλα καλά, ε, γιατί είναι πολύ σημαντικό το ότι δεν έχουμε αξιοποιήσει στο έπακρο το δυναμικό του ευρωπαϊκού εξαμήνου. Οι μακροοικονομικές ανισορροπίες θα πρέπει να λαμβάνονται πιο σοβαρά υπόψη, έχουν πιο ασθενή νομική βάση, ωστόσο θα πρέπει να λαμβάνονται πιο σοβαρά υπόψη, επαναλαμβάνω. Και είναι θέμα να έχει κανεί τεράστιο πλεόνασμα τρεχούσων συναλλαγών. Εξίσου μεγάλο θέμα όπως είναι το θέμα του ελλείμματο και του χρέους. Θα πρέπει ε, να μπορούμε να έχουμε αθρηστική ε, δημοσιονομική ε, παρουσία Αρχικά ο Επίτροπος είχε ζητήσει το ξαναχτίσιμο ενός ε, δημοσιονομικού μπάφερ, ενός μαξιλαριού και τώρα πάμε σε επεκτατικές ε, ε, δημοσιονομικές πολιτικές. Όλα αυτά όμως σχετίζονται με τις ατομικές διαπραγματεύσεις. Το σημαντικό είναι να έχει αθρηστικά η ζώνη του ευρώ τη δυνατότητα να λειτουργήσει αντικυκλικά. Πολλά πρέπει να βελτιώσουμε σε αυτό το πεδίο. Θα πρέπει να έχουμε πιο απλούς κανόνες και περιμένουμε το νέο κύκλο μεταρρυθμίσεων που έχει ανακαινώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα επόμενα χρόνια και κάτι το πολύ σημαντικό για μένα είναι ότι χρειαζόμαστε μια πιο ισχυρή ε, η δυνατότητα σε επίπεδο φορολογικών και δημοσιονομικών, αν θέλετε. Δεν θα έχουμε την βελτίωση του συντονισμού μόνο μέσω εθνικών πολιτικών. Το αληθινό εργαλείο είναι να έχουμε ισχυρότερη δημοσιονομική δυνατότητα και αυτό ισχύει και για τις επενδύσεις και για τους άλλους τομείς. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε αυτό το εργαλείο για τη σταθεροποίηση και αυτό είναι απαραίτητο για την ολοκλήρωση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης. Η Μαριάν Τάισεν είπε κάτι που με βρίσκει απολύτως σύμφωνο. Θα πρέπει να κάνουμε περισσότερο για την καλύτερη συμπερίληψη του εργασιακού και κοινωνικού πυλώνα. Η αυτή η Επιτροπή έκανε πολλά προς αυτήν την κατεύθυνση, αλλά πρέπει να κάνουμε ακόμα περισσότερα για να εφαρμόσουμε και να υλοποιήσουμε τον εργασιακό πυλώνα. Πολλοί συνάδελφοι αναφέρθηκαν στον εκδημοκρατισμό της διαδικασίας και αυτό είναι σημαντικό. Είναι μια πρόκληση βεβαίως, γιατί η συγκεκριμένη διάσκεψη δεν βασίζεται σε σταθμισμένο βάρος των κρατών μελών και των πληθυσμών, δεν μπορούμε να ε, ψηφίσουμε με δεσμευτικό τρόπο, δεν υπάρχει και νομική βάση. Όμω, ανακοινώνουμε διάλογο και συνεργασία μεταξύ Εθνικών Κοινοβουλίων και, σε Ευρωπαϊκού, ε, και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και σε επίπεδο ολομέλεια και σε επίπεδο πολιτικών οικογενειών. Όλα αυτά είναι απαραίτητη βάση για να χτίσουμε μια κοινή κουλτούρα όπου όλοι θα βρισκόμαστε στην ίδια βάρκα, στο ίδιο πλοίο και η ιδιοκτησία υπευθυνότητα σημαίνει η ε, δυνατότητα συντονισμού σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο σημαίνει να βρίσκουμε προτεραιότητες, να κατευθύνουμε ε, μια ευρωπαϊκή διαδικασία διαμέσου των διαφόρων επιμέρους εθνικών διαδικασιών. Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά. Σας ευχαριστώ για τη συνεισφορά σας. Με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον θα παρακολουθήσω την αυριανή συζήτηση όπου θα αναπτύξουμε με ακόμα πιο ζωντανό τρόπο όλα αυτά τα θέματα που μας απασχολούν για να καλλιεργήσουμε το διάλογο και να δώσουμε δημοκρατική όθηση στην, στο Ευρωπαϊκό Εξάμεινο και στην ολοκλήρωση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης. Μιλώντας άλλωστε και για το κίνδυνο της βραδίας ανάπτυξης και της βραδίας ανάκαμψης. Σας ευχαριστώ όλους. Δίνω το λόγο στη Συμπρόεδρο για τις ε, καταληκτικές της παρατηρήσεις. Ευχαριστώ. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Ε, πρότιμο να μιλήσω τη μητρική μου γλώσσα για να κλείσω. Στα ρουμανικά θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πολύ όλους σας, όλους τους συναδελφούς από τα Εθνικά Κοινοβούλια, όλους τους Ευρωβουλευτές για την παρουσία σας εδώ ανεξαρτήτως ε, πολιτικής ε, παράταξης και οικογένειας, δεξί, αριστερή. Βεβαίως, πολλοί είμαστε δυσαρεστημένοι, εκφράζουμε την απογοήτευσή μας, αλλά ε, όλα αυτά μπορούμε να τα ξεπεράσουμε. Και στη δική μου χώρα ακούμε διάφορα δυσάρεστα που συμβαίνουν. Ε, πάντως, όταν υπάρχει καλή θέληση, συνεργασία ε, όλα τα προβλήματα ε, μπορούν να ξεπεραστούν. Η Ρουμανική Προεδρία φυσικά ε, θέλει να συνεχίσει να εργάζεται σε πολλά από τα θέματα που εκκρεμούν για να προχωρήσουν να και ολοκληρωθούν. Σε, αυτό, σε αυτά ανήκουν και το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο και οι επενδύσεις και τα μεγάλα έργα. Και αυτά θα πρέπει να ε, υλοποιούνται σε όλα τα κράτη-μέλη. Σας ευχαριστώ και πάλι για τη συζήτηση αυτή, για την παρουσία σας, για τα ενδιαφέροντα που ε, ακούσαμε και ελπίζω να τα ξαναπούμε και αύριο με νέες δυνάμεις για να συνεχίσουμε τη συζήτηση αυτή. Ευχαριστώ πολύ. Thank you. Just a technical note now. Ένα τεχνικό τώρα. Έχουμε τρεις παράλληλες συνεδριάσεις. Ε, οικονομική στην αίθουσα PHS 3 σε 50 που είναι ακριβώς απέναντι από την Ολομέλεια. Ε, στο Γιάν 4 ε, η άλλη συνεδρίαση και ο προπολογισμό ε, Γιάν 6-2. 4Q1 είναι τα κοινωνικά. Ναι.